Buongiorno a tutti. Καλησπέρα σας. Θα κάνουμε έλεγχο των συσκευών μας. C'era l'aereo in ritardo. Vediamo. Mm? Il voto è aperto. Άρχεται η ψηφοφορία. Έλεγχος των συσκευών. Άρχεται Άρχεται η ψηφοφορία, ή αρχίζει τουλάχιστον, μέχρι θα το καθίσουν όλοι. Κυρίως ο κύριος Γκέρενς. Hai votato Strifel tu che devi prendere l'aereo, sì? Dare la parola a Guillaume. Bene, ok. Diamo subito la parola, chiede l'onorevole Guillaume, prego. Το λόγο ζητά ο κύριος Περιμένω την ηλεκτρονική μου κάρτα, θα καταθάσει ανα πάσα στιγμή. Αν μου επιτρέπετε στο μεταξύ να ψηφίζω διανατάσταση της χειρός. Ναι. Οκ. Chiuso, λοιπόν, Τέλος ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε κανονικά τώρα το σχέδιο για τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γρυλανδίας και Βασιλείου της Δανίας. 28. Ε, Ποιος είναι υπέρ. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεν έχετε καμία εμπιστοσύνη. Ε. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έρχεται η ψηφοφορία. Il voto Τέλος ψηφοφορίας. Αγκρίνεται, όντως. Έχατε δίκιο. Συνεχίζουμε. Ψηφίζουμε ομάδων, αν δεν έχετε αντίρρηση, τις τροπολογίες 29 έως 34. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Μήπως θέλει κανείς ηλεκτρονικό έλεγχο πάλι? Όχι κανείς. Εγκρίνονται άλλωστε. Τροπολογία 35. Ψηφίζουμε και εδώ 35 ως 40 και μετά 26 και 27, όλες μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Σας ορκίζομαι ότι εγκρίνονται. Τροπολογία 36. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. 37 τώρα, τροπολογία 37. Και εδώ θα τις ψηφίσουμε μαζί. Αμα έτσι θα τελειώσουμε πολύ γρήγορα. Δεν μου δίνετε καν την ικανοποίηση να προεδρεύσω λίγο σε ψηφοφορίες. Καλά, 37 και έως 42 Μαζί παρακαλώ. Ποιος, ποιο, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον εγκρίνονται. Ή μήπως κάνω λάθος. Όχι, εγκρίνονται. Και πάλι ομαδών τις υπόλοιπες τροπολογίες. Με εξαίρεση την 20. Την 20 θα την ψηφίσουμε ξεχωριστά. Ωραία, ποιος είναι υπέρ της 20. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Γιατί ψήφισα τρεις φορές. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα θα ψηφίσουμε από κοινού τις 21 έως την 25. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Θα ψηφίσουμε τώρα την ούτως τραποποιηθήσα έκθεση. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ποιος είναι υπέρ? Ή μάλλον ηλεκτρονικά, λέει η πρόεδρος. Όχι, ηλεκτρονικά. Διανατάσεις χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το σχέδιο έκθεσης με τις τροπολογίες. Τώρα θα ψηφίσουμε την πρόταση ψηφίσματος, νομοθετικού ψηφίσματος, ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά λοιπόν το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος άρχεται η ψηφοφορία. Ποιος είναι η λέει πρόεδρος. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ψηφί. Τι ωραία, όλοι συμφωνούμε. Υπάρχουν σχόλια. Ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο ψηφίσματος για τον υποσυτισμό των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ψηφοφορία εδώ είναι απλούστατη γιατί δεν έχουν υποβληθεί τροπολογίες. Ψηφίζουμε κατευθείαν και ηλεκτρονικά την πρόταση ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Υπέρλυ, πρόεδρος κατά αποχές εγκρίνεται, αν και η δική μου κάρτα δεν λειτουργεί από ό,τι φαίνεται. Και εγώ ψήφισα υπέρ. Ούτε η δική σας ε, λειτουργεί. Ούτε εσείς ψηφίσατε. Επανάληψη της ψηφοφορίας. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται ομόφωνα τι είπα προηγουμένως να διαβάσω αυτό το κείμενο πρόκειται για μια οριζόντια τροπολογία που αν εγκριθεί θα αντικατασταθεί ο όρος υποσυτισμός ε, από το ε, Από το malnutrition, από το denutrition. Αν απορριφθεί, οι υπόλοιπες οι θα καταπέσουν, οπότε θα παραμείνουμε στον όρο υποσυτισμός. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρχιτη ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 14 ψήφους υπέρ 10 κατά. Τροπολογία 8. Δεν είμαι εμπειρογνώμων, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει το under nutrition, under nourished λέμε στα αγγλικά, για τον υποσυτισμό. Malnourished και under-nourished εκεί είναι η διαφορά. δεν denutrition, είναι συναφής οι όροι. Στα ελληνικά υποσυτισμός λέμε. Τώρα δεν ξέρω, ίσως πρέπει να παραπέμψουμε το θέμα στους γλωσσομαθείς νομικούς για να μας πούν ποιος είναι ο πιο δόκιμος όρος. Κύριε Κάσμα, μπορούμε να συνεχίσουμε. Έχετε δίκιο. Ε, συνεχίζουμε. Τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Προβάτο. Εγκρίνεται. 15, 16, 21, 22 και 23 μαζί. Γιατί η τροπολογία 17 και 20 έχουν καταπέσει. Ποιος είναι υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνονται. Πολύ ωραία. Έχουμε μία ακόμη ομάδα τροπολογιών. Όχι, ξεχωριστά. Τη τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά άποχες Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 4. Ε, η κυρία ζητάει έλεγχο, αλλά είναι μειοψηφία. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονικά. Προτιμά ηλεκτρονικά εδώ ο κύριος. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Υπέρ. πρέπει να ψηφίσουμε δύο φορές και με τους δύο τρόπους. Πρώτα, διανατάσσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερη ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά, αποχές. Τέλος της ψηφοφορίας και εγκρίνεται ομόφωνα μάλιστα. Εντάξει, ακόμη και τις ψηφοφορίες λίγη χαρά κακό δεν κάνει. Είμαστε συνήθως τόσο κατηφείς όλοι. Περνάμε στο σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα την εξάλληψη των βασανιστήριων στον κόσμο. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ, ή να ψηφίσουμε συνολικά τις τροπολογίες. Όχι, ξεχωριστά. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τέσσερα. Ή θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Αφού εσείς ψηφίσετε κατά, σας έδωσα δίκιο. Είπα απορρίπτεται και θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Κύριε Κορτές. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 5 καταπίπτει. Προχωράμε στην 6. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κατά τη γνώμη μου απορρίπτεται. Αλλά αν θέλετε να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά, καμία αντίρρηση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε με 16 ψήφους κατά και 8 υπέρ. Προφορική τροπολογία. ή μάλλον τροπολογία 2 διορθώνει η πρόεδρος. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ο τροπολογία 8 καταπίπτει, περνάμε στην τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10, υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο γνωμοδότησης, όπως έχει τροποποιηθεί, με τα χέρια, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται ομόφωνα. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία των τροπολογιών 1 έως 9 Ποιος είναι υπέρ. Κάποιος διαφωνεί. Εσείς έχετε δίκιο. Λοιπόν, τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά, αποχές. εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές Ωραία, εγκρίνεται. Μόνο ένα είναι κατά. Έξι. Έχετε δίκιο. Γιατί να τι ψηφίσουμε μαζί. Δίκιο έχει ο άνθρωπο, είναι κατά. Μην με μπερδεύετε. Ποιο είναι υπέρ. Ή εσεί θέλετε, εσεί ζητήσατε να τι ψηφίσουμε μαζί. Μέχρι το τέλο. Ωραία. Όλε οι υπόλοιπε υπέρ, κατά, αποχέ. Εγκρίνονται. Χειροκρότημα για σας. Και τώρα λίγη σοβαρότητα. Αν γίνεται. Ψηφίζουμε την ε, γνωμαδότηση όπως έχει τροποποιηθεί. Υπέρ, κατά, αποχές. Θέλετε και ηλεκτρονικό έλεγχο. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Πρέπει να λέω κάθε φορά άρχεται η ψηφοφορία. Μάλιστα. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν κυρίες και κύριοι. Υπέρ, κατά, αποχές. Τέλος της ψηφοφορίας. Μπράβο, συγχαρητήρια. 23 υπέρ, 1 κατά. Μα τι μυστική ψηφοφορία, κοιτάξτε. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τις ψηφοφορίες, αγαπητοί συνάδελφοι. Πώς τα πήγα, τα κατάφερα, ευχαριστώ, καλή μου. Adesso lei felicita la venuta di due persone che sono Un momento, eh, Goerens vuol prendere la parola. Eh, merci, Madame la Présidente. Ok, κύριος Goerens, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το είχα επισημάνει και σε προηγούμενη συνεδρίαση. Ουδέποτε δεν κατάλαβα γιατί ψηφίζουμε πρώτα διανατάσεις τη χειρό και έχουμε και δεύτερη ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Είναι τελείως παράλογο. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν θα έπρεπε να το ομολογήσω, αλλά έτσι αποφάσισαν οι συντονιστές. Οι συντονιστές το αποφάσισαν. Δική του απόφαση είναι να ψηφίζουμε δύο φορές. Μα εγώ συντονιστή είμαι. Δεν θυμάμαι να είχα δώσει τη σύμφωνη γνώμη μου για τέτοια χαζομάρα. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ τον Αντιπρόεδρο του, της Μεξικανικής Γερουσίας, τον κύριο Ρενέ Ζωζέα Ισπούρο Τόρες και τον κύριο Αρτούρο Γκαρίτα, που είναι Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Μεξικανικής Γερουσίας. Καλώς ήρθατε. Bene, adesso continuiamo Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά τις ψηφοφορίες ε, θα ακούσουμε την παρουσίαση εκ μέρους του κυρίου Γκέρενς της έκθεσης, του σχεδίου έκθεσης του με θέμα τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Συγχαρητήρια κύριε Γκέρες, εργάζεστε άοπνα πραγματικά. Είστε πολύ εργατικός. Έχετε το λόγο. Ε, ε, ε, κύριε Γκέρενς, έχετε το λόγο. Μας μιλήσετε για την σχετική έκθεση, την συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη. Θέλετε να μιλήσετε. Αλλιώς ε, να δώσουμε το λόγο σε κάποιον άλλον. Κυρία Πρόεδρε, την περσμένη φορά ξέρετε ήμασταν μόνο τρεις, γι' αυτό διστάζω. Αν μαζευτούμε περισσότεροι να ξεκινήσω. Λοιπόν, εντάχει. Έχω ήδη σημειώσει ότι στην αρχή τη Κυρία έχουμε πει ουσιαστικά τα πάντα. Εγώ εστιάζομαι σε κάποιες προτεραιότητες, σε συγκεκριμένε προτεραιότητες. Το βασικό μήνυμα είναι το εξή. Το δεύτερο μέρος της παρουσίασης μου αφορά την μέθοδο. Ε, μετά τη δεν είναι δυνατόν όμως Πρόεδρος. Όποιος δεν ενδιαφέρεται να βγει παρακαλώ. Κύριε Όσον αφορά την μέθοδο, η κριτική μου ενάντια της Κομισιόν είναι η εξής. Περιμένουμε ανακοίνωση της Κομισιόν με την οποία θα δεσμευόταν το σύνολο της Κομισιόν. Τώρα έχουμε ένα έγγραφο εργασία το οποίο δεσμεύει μόνο την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αυτό είναι το βασικό πολιτικό πρόβλημα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε. Γιατί, διότι πού κρίνεται το θέμα, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ δύο συγκεκριμένων πολιτικών. Δεν θα προκρίνει λύση η αρμόδια διευθύνση. Το θέμα είναι λοιπόν ποιος θα είναι αρμόδιος να κρίνει το ζήτημα στην περίπτωση σύγκρουσης. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι ο πρόεδρος ο ίδιος της Κομισιόν. Στο υψηλότερο δηλαδή επίπεδο. Και το ίδιο ισχύει για τα κράτη-μέλη. Για όσους έχουν αναλάβει εκτελεστικούς ρόλους σε εθνικό επίπεδο, θα λέω ότι γνωρίζουν το θέμα, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Δηλαδή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αν δεν ξέρουμε ποιο όργανο διαθέτει επαρκείς εξουσίες και αρμοδιότητες για να μπορεί να προκρίνει λύσεις σε τέτοιου είδους συγκρούσεις. Στο σχέδιο ψηφίσματος επιμένω να συμπεριληφθεί ο στόχος της ε, συμβερότητας των πολιτικών στο πλαίσιο μετά το 2015 ως προς το καθεστώς του εγγράφου, σας τα είπα ήδη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πλευρά του και ως προς την μέθοδο συγκεκριμένα έχει κάθε λόγο να δημιουργήσει μικτές επιτροπές έτσι ώστε και εμείς να μπορούμε να εκπονούμε γνωμοδοτήσεις προσαρμοσμένε απαιτήσει τη της πολιτικής ανάπτυξης. Όσον αφορά του τομεί προτεραιότητε, αναφέρω μετανάστευση, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε επιπτώσει τη της ΚΑΠ, της κοινή αγροτικής πολιτικής, των τομέα τη ανάπτυξης, πιστεύω ότι επαναλαμβάνω εδώ πιστά τις ανησυχίες των συναδέλφων, και αναφέρομαι και σε άλλα ζητήματα όπως ε, τα μεγάλα έργα υποδομών στον τομέα της ενέργειας που έχουν επιπτώσει στην εφορική ανάπτυξη. Αναφέρουμε και στην Ελία. Σε αυτά θα περιοριστώ κυρία Πρόεδρε, Εισαγωγικό και αναμένω σχόλια. Ευχαριστώ. Υπάρχει κανείς που θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Μίτσελ. Ως και όδης συζητητής ε, Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι υποστηρίζω την προσέγγιση του Τσάρλς σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία ανέφερε. Πρόκειται για ένα πολύ βασικό εργαλείο της Επιτροπής μας και νομίζω ότι ο Τσαρλ έχει επιδείξει κάποια σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σε ό,τι αφορά ε, την συνεκτικότητα της πολιτικής, σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή ατζέντα. Ήμουνα εισηγητή σε ό,τι αφορά το συντονισμό των δωρετών, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή βοήθεια. Πολλά λοιπόν ε, τέτοια θέματα μπορούμε να τα ε, αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο και χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είτε πρόκειται για την ε, εξοικονόμηση πόρων, είτε πρόκειται για την ε, συνεκτικότητα των πολιτικών. Καλωσορίζω αυτά που είπε ο Τσάρλς μόλις για τη συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής και σε θέματα συνεκτικότητας ε, της πολιτικής. Γεωργία, εμπόριο, υγεία, αλληλεία, περιβάλλον. Αν και οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Γεωργίας μου λένε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ακαθόδη όσο στο παρελθόν, θεωρώ παρόλα αυτά ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την διάδραση μεταξύ των πολιτικών αυτών και σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια αλλά και μεταξύ τους. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να το θίξουμε το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την ευκαιρία της έκθεσης ε, του Τσάρλς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να θίξουμε δηλαδή την πολιτική βούληση για την αναπτυξιακή βοήθεια. Υποστηρίζω επίσης αυτά που είπε ο Τσάρλς για την πρόταση να συμπεριληφθεί η συνεκτικότητα της πολιτικής την φάση και στο πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2015. Αν θέλουμε να σταθεί με επιτυχία και αυτή η νέα περίοδος θα πρέπει να κοιτάξουμε τι προβλήματα συντονισμού πολιτικής δωρητών είχαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Ανεξάρτητα από την τεράστια επιτυχία των NDG Χρειάζεται προσπάθεια για τον συντονισμό από χώρα σε χώρα και από οργάνωση σε οργάνωση. Και νομίζω ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συνεκτικότητα αν θέλουμε να πετύχουμε μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε λοιπόν τον συνάδελφο κύριο Γκέρενς για την έκθεσή του και υποστηρίζω πολλά από τα συγκεκριμένα στοιχεία, πολλά των οποίων ενδεχομένω να προκαλέσουν προβλήματα σε άλλε επιτροπέ, αλλά εμεί πρέπει να τα προωθήσουμε, γιατί αν το κάνουμε εμεί δεν θα το πράξει κανεί άλλο. Σα ευχαριστώ και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Νέιζερ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, τον κύριο Γκέρεντ, επειδή η έκθεσή του ήταν σύντομη, συνοπτική, αλλά και πλούσια σε περιεχόμενο. Και θέτει το θέμα επιτάπητος. Στην έκθεση ζητείται ένας μηχανισμός προστασίας, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται στα χέρια του Προέδρου της Επιτροπής. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό ως ε, σύστημα για να μπορούν έτσι να επιλύονται ενδεχόμενα προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται και στην περίοδο μετά το 2015 για τους αναπτυξιακούς στόχους. Να συμπεριληφθεί επίσης αυτός ε, ε, όρος συνοχής για να μην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στη γεωργία και σε άλλους κλάδους των αναπτυσσόμενων χωρών. Θέλουμε να, να καθίσετε σαφές και στην έκθεση ότι θα συνεχίσει να διδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημαντικό ρόλο για να υπάρχει ακριβώς αυτή η συνεκτικότητα. Και αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε έναν ανεξάρτητο ελεκτικό μηχανισμό, τότε οι πολίτες μας, αλλά και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, θα έχουν την ευκαιρία όπου δει να δίνουν πρόσβαση σε εμά στο Κοινοβούλιο σε τέτοια θέματα για να μπορέσουμε να τα επιληφθούμε αυτών. Θεωρώ ότι είναι σαφή τα προβληματικά σημεία τα οποία εντοπίζονται μετανάστευση, εμπόριο, γεωργία, αλληλεία και η αλλαγή του κλίματος. Και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερο σημαντικό για μας το θέμα των υποδομών και της ενέργειας, προκειμένου να κοιτάξουμε τα πιο μικρά διαρθωτικά έργα. Καλή έκθεση. Από δική μας πλευράς δεν θα υπάρξουν ούτε προσθήκες ούτε τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ε, Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριο Φροντίνη Γκάσπερ. Είναι εδώ, όχι. Όχι. Καλή αργά παρά ποτέ. Να περιμένουμε ένα λεπτό να κάτσει. Ο κύριος Φραντίνη Γκάσπερ, καλώς ορίσατε. Μπορεί να μην έχετε ακούσει τίποτα, αλλά θα πρέπει να μπείτε κατευθείαν στο θέμα. Ναι, ναι, ναι, έχουμε, έχουμε εμπιστοσύνη. Thank you. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και λυπάμαι που καθυστέρησα. Εγώ νόμιζα ότι δεν είχα καθυστερήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει μάλλον ήρθα λίγο αργότερα. σα ευχαριστώ που μου δίνετε και την ευκαιρία να σχολιάσω την έκθεση. Και αυτά που μου είπαν για τη συζήτηση που έλαβε χώρα. Να πω ότι είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με την καλή υποδοχή της δικής μας ε, Έκθεση εδώ στην Επιτροπή σας το Νοέμβριο, όταν τη συζητήσαμε. Επίσης έγινε καλή συζήτηση στο, Ευρωπαϊκό, Συμβούλιο ε, και αποτυπώνεται αυτά και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Καλώς ορίζουμε επίσης τον πολύ επικοδομητικό ύφο της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλώς ορίζουμε και τις ε, πολύ άριθμες προτάσεις τις οποίες κάνατε προκειμένου να καταστεί το PCD ένα πιο λειτουργικό εργαλείο, το οποίο ασφαλώς αποτελεί και αυτό σκοπό μας και ασφαλώς αυτό επιδιώκουμε. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερως που μπορούμε να υπολογίζουμε στην συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλωσορίζουμε επίσης ε, το πεδίο εφαρμογή των ε, συστάσεων που έχουν διατυπωθεί επιμένοντα τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάποιε από τι προτάσει ήταν ασφαλώ ζητήματα τα οποία και εμείς είχαμε τονίσει στη δική μας έκθεση. Προκειμένου τώρα να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος για το μορφότυπο. Το παρουσιάσαμε αυτό ως ένα έγγραφο εργασίας γιατί είναι ένα εργαλείο υποβολής αναφορών που εξετάζει και τις δραστηριότητε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλων των κρατών μελών. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το εργαλείο της, ε, των αναφορών. Αλλά αυτό χρησιμοποιείται και για την ε, επικοινωνιακή διάσταση και για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής. Αλλά βλέπετε ότι είναι καλός ο μορφότυπος της έκθεσης της αναφοράς. Δεν αποτέλεσε πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις στο Συμβούλιο Υιοθετήθηκαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά και την έκθεση και έγιναν συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή διάσταση. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια. Παρουσιάσαμε και το θέμα αυτό στις Ευρωπαϊκές ημέρες ανάπτυξης, προσπαθούμε να το παρουσιάσουμε και στα διάφορα κρατημέλη, καταβάλουμε προσπάθεια να μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες, να είναι πιο εύκολη η ανάγνωση από το κοινό. σε ό,τι αφορά την περίοδο μετά το 2015 και τις συστάσεις που έγιναν. Νομίζω ότι εδώ συμφωνούμε στις αντρές γραμμές. Βλέπουμε ότι αυτό αποτελεί μία ευκαιρία προκειμένου αυτή η συνοχή της ανεπτυξιακής πολιτικής να τεθεί σε διεθνές επίπεδο. Το κάναμε αυτό λοιπόν, συντονίσαμε την πολιτική αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πάρα πολύ ωφέλιμο, αλλά εξίσου ωφέλιμο να μεταφερθεί αυτό ως αρχή στη διεθνή κοινότητα εκτός Ευρώπης, όπου συχνά η αρχή αυτή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής είναι άγνωστη. Νομίζουμε λοιπόν ότι οι συζητήσει για την περίοδο μετά το 2015 αποτελούν μια καλή ευκαιρία για να το πράξουμε αυτό. Πώς θα αποτυπωθεί αυτό. Θέλουμε να αποτυπώνεται το PCD, η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής στο επόμενο πλαίσιο. Αυτό θα εξαρτηθεί και από το πώς θα δημοφιλωθεί το ίδιο το πλαίσιο θα πρέπει να βρούμε τη σωστή θέση στις συζητήσεις σε ό,τι αφορά και την εφαρμογή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής. Και εδώ θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο σκέλη στην εφαρμογή. Χρηματοδότηση αφενός και πολιτικές αφετέρου. Πολιτικές λοιπόν σε αυτό το σημείο εντάσσεται και το PCD, η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σχόλια που γίνονται στην έκθεση για το εμπόριο, θεωρούμε ότι η γλώσσα θα μπορούσε να είναι και λίγο πιο θετική, πιο αισιόδοξη. Υπογραμμίζονται κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά το εμπόριο, αλλά υπάρχουν και πολύ σημαντικά θέματα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Υπό τον όρο φυσικά ότι υπάρχουν καλές εγχώριες πολιτικές. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρώτος τέτοιος εταίρος σε παγκόσμιο επίπεδο, νομίζω ότι μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο της σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη τώρα, σε ό,τι αφορά τα σχόλια της κοινής αγροτικής πολιτικής και την ανάγκη να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος. Προσπαθούμε όχι μόνο για την κοινή γεωργική πολιτική, αλλά για όλες τις πρωτοβουλίες της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο να δούμε πώς μπορεί να προσμετρηθεί και να υπολογιστεί λοιπόν ο αντικτύπος στις τρίτες χώρες. Αυτό είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά σας προειδοποιώ ότι οι ποσοτικές αξιολογήσεις για κάποιες χώρες, ιδιαίτερα σε θέματα γεωργία, έχουμε πρόβλημα πρόσβαση στα δεδομένα. Δεν έχουμε πάντα τα απαραίτητα στοιχεία για να κάνουμε τις αξιολογήσεις αυτές, τις εκτιμήσει αυτέ. Άρα εδώ βάζω να. Ε, ερωτηματικό, δεν είναι θαυμαστικό σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, την ενέργεια, την αλληλεία, την κλιματική αλλαγή. Θεωρώ ότι είναι προτεραιότητες κλειδί, γι' αυτό συμφωνούμε. Εδώ λοιπόν προσπαθούμε για όλα αυτά να τα εντάξουμε στον προγραμματισμό μας. Είμαστε σε φάση ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα του συντονισμού, Είναι κοινό το καθήκον μας και με την Υπηρεσία Εξωτερική δράση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτιθέμεθα να συνεργαστούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής θα εφαρμοστεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Με κύριο Γκέρεντς. Ευχαριστώ επί της ουσίας συμφωνούμε για τα περισσότερα τουλάχιστον θέματα, αλλά στο θέμα της ε, επιδητησίας αυτής θα ήθελα να πούμε δύο κουβέρες παραπάνω. Από την αρχή είχαμε ζητήσει από την Κομισιόν να εκδώσει, είπα, ανακοίνωση με την οποία να δεσμεύεται το σύνολο των επιτρόπων. Δεν ξέρω αν έφτασε το θυμά μας ως τον Μπαρόζο. Μπορεί να μην του καίγεται καρφάκι δεν το αποκλείω αυτό το γεγονός, εν πάση περιπτώσει, όταν έρθει η ώρα να ψηφίσουμε επί της εκθέσεως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει θέση και να μας πει τι συνέχεια θέλει να δώσει στο αίτημά μας. Απαιτώ η Κομισιόν να τοποθετηθεί επί του αιτήματός μας. Θέλω να ξέρω τη γνώμη όχι μόνο του Πίλμπαξ, αλλά όλων των επιτρόπων, αρχίζοντα από τον πρόεδρο τη Κομισιόν. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα ουσία. Μπορούμε να γράφουμε σχολικέ εκθέσει ε, κάθε εξάμεινο, κάθε χρόνο, αν θέλετε, αλλά αν δεν σημειωθεί πρόοδο στο συγκεκριμένο θέμα τη επίλυση αυτών των ε, συγκρούσεων, στην περίπτωση που υπάρχουν βεβαίω συγκρούσει, τότε δεν έχουμε κάνει τίποτα. Γι' αυτό και αναμένω στο ακουστικό μου ως προς το αίτημα το οποίο θα επαναλάβω ενώπιον της Ολομελίας δεν μπορώ να το πω πιο συγκεκριμένα τώρα όσον αφορά άλλες συστάσεις θα το δούμε στην Ολομελία να δούμε πώς θα τοποθετηθούμε και μετά θα, προ... θα διατυπώσουμε συστάσεις σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Οπότε θα μιλήσω πλέον ενώπιον των συντονιστών πιο συγκεκριμένα και σε, επί αυτού που είπε και ο συνάδελφος Μίτσελ για να δούμε λοιπόν πώς θα συνεργαστούμε με τα εθνικά κοινοβούλια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είμαι εν γέννη αρκετά ικανοποιημένο από τη συζήτηση διότι περιοριστήκαμε επί δύο συγκεκριμένων πτυχών πολύ σημαντικών πτυχών χωρίς να παραλαμβάνουμε τα γνωστά. Και κλείνω λέγοντας ότι υιοθετούμε μια προσέγγιση στο πλαίσιο της οποίας δημιουργούμε μια επιτροπή, ορίζουμε εισηγητή, εντοπίζουμε τους τομείς στους οποίους ενδέχεται να εμφανιστούν να προκύψουν συγκρούσεις Και κάποια στιγμή κάποιοι θα μα πούνε να φτιάξουμε μια task force κλπ. Λοιπόν, αυτά όμω δεν μα οδηγούν πουθενά. Να πάρουμε μια απόφαση για τη μέθοδο, για μια συγκεκριμένη μέθοδο. Εμεί δεν θα το παρατήσουμε το θέμα. Ε, πιστεύω ότι δεν σπαταλήσαμε το χρόνο μα ε, κάνοντα τι κάναμε. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για το σχέδιο έκθεση. Ε, λίγη στις 29 Ιανουαρίου, το μεσημέρι. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξής μας είναι η παρουσίαση της μελέτης ε, με θέμα το μαλλί και τους οικονομικούς παράγοντες ε, πίσω από την κρίση. Θα δώσω το λόγο αμέσως στην κυρία Φραντσέσκα Μπαστάλη για 20 λεπτά είναι η συντάκτρια της μελέτης. My name is Καλησπέρα σας, ε, Φρανσίσκα Μαστάλη ονομάζομαι και είμαι ερευνήτρια στο ε, Ινστιτούτο του Λονδίνου και σας, ε, θα σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά μια μελέτη για τους οικονομικούς παράγοντες πίσω από τις κρίσεις του Μάλι. Έχετε νομίζω τη μελέτη Μπροστά σας έχετε τη διαφάνεια. Η... Την ε, μελέτη την ανέθεσε σε εμά το Κοινοβούλιο. Μα ζήτησε να δώσουμε μια επισκόπηση της οικονομίας και τις ε, πρόσφατες τάσεις μέχρι το 2012 που οδήγησαν στην κρίση. Και κάποιες πληροφορίες για το τι συνέβη μετά το 2012 και κάποιες συστάσεις ε, βάσει των αναλυσεών μας. Αυτή τη γραμμή λοιπόν θα ακολουθήσω και στην παρουσίασή μου σήμερα. Θα είμαι σύντομη στην παρουσίασή μου. Θα βρείτε πιο απλές πληροφορίες αν θέλετε σε έγγραφη μορφή. Να σας παρουσιάσω λοιπόν κάποια από τα απορίσματα σε ό,τι αφορά τις τάσεις και τις πολιτικές, τις οικονομικές πολιτικές μέχρι το 12. Μετά θα κοιτάξουμε κάποια στοιχεία και τάσεις για την ένδυα, την ανισότητα και τις κοινωνικές πολιτικές. Θα εντοπίσουμε τις βασικές προκλήσεις στην εφαρμογή πολιτικής. Θα σας δώσουμε μια επισκόμιση του ρόλου των διεθνών και περιφερειακών φορέων. Θα κοιτάξουμε τις εξελίξεις μετά την, ε, το ξέσπασμα της κρίσης και... Στη συνέχεια θα δούμε τις συστάσεις σε ό,τι αφορά το ΟΜΑΛΗ και την ε, οικονομία του Μαλή. Σε ό,τι αφορά την οικονομία, το γενικό συμπέρασμα και το γενικό πόρισμα της μελέτης είναι ότι καταδεικνύεται ότι μακροοικονομικά το Μαλή τα πηγαίνει καλά. Συνάδει με τα κριτήρια εκείνα και τους όρους εκείνους που θέτουν οι διεθνείς ε, χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και οι περιφερειακοί σχετικοί οργανισμοί τα τελευταία χρόνια. Εξετάζοντας την οικονομική ανάπτυξη, εν γέννη θεωρείται ότι είναι καλό το κατά, το κατά ε, ΑΕΠ του Μαλή. Κατά 4,9% αναπτυχτική οικονομία τα τελευταία χρόνια από το 2007-2010 και όπως φαντάζεστε αυτό επηρεάστηκε από τη ξέσπασμα της βίας το 2012. Η ανάπτυξη χρηματοδοτείται κυρίως από την γεωργία και από τον τουρισμό, τις τηλεπικοινωνίες, ενώ ο δευτερογενής τομέας έχει σημειώσει πτώση τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, υπάρχουν δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη αυτή, που πιστεύω ότι ε, αξίζει να τα επισημάνουμε. Καταρχάς, κοιτώντας την κατακεφαλή ανάπτυξη του ΑΕΠ, είναι πολύ αργή η κατακεφαλή ανάπτυξη του ΑΕΠ. Στην ίδια λοιπόν περίοδο μιλάμε για 1,4% ανάπτυξη κατακεφαλή. Αυτό οφείλεται εν μέρη στην μεγάλη αύξηση του πληθυσμού. Ένα δεύτερο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η ανάπτυξη δεν μεταφράστηκε σε αύξηση της απασχολησιμότητας. Μάλιστα αυξήθηκε ελαφριά η ανεργία και όπου δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας ήταν στον ανεπίσημο τομέα. Κοιτώντας τα δημοσιονομικά τώρα, θετικές οι αξιολογήσεις και πάλι εν γέννη υποδεικνύουν ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές είναι ιδέουσες και έχουν γίνει οι κατάλληλες προσπάθειες για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Έχουν σημειωθεί σωστές ε, πρόοδοι, αύξηση των κυβερνητικών εσόδων, αυτό κατά μεγάλο βαθμό από αύξηση της φορολογίας, θετικό αποτέλεσμα και οι δαπάνες έχουν προσαρμοστεί στις τάσεις των προσόδων. Αυτό ασφαλώς αποτελεί ένα μέτρο ε, σωστής δημοσιονομικής πολιτικής. Το 2008, για παράδειγμα, όταν μετά την κρίση το, λόγω της τιμής των τροφίμων ε, μειώθηκαν τα έσοδα, μειώθηκαν και οι δαπάνες. Ενώ γενικά προστατεύονται οι κοινωνικές δαπάνες στην υγεία, στην παιδεία. Αυτά τα γενικά αποτελέσματα αποτελούν ενδείξεις και τμήματα μιας καλής δημοσιονομικής πολιτικής και μιας σωστή φορολογικής πολιτικής και ε, κρατικών δαπανών. Εκ παραλλήλου, εξετάζοντας τον τομέα των εξαγωγών και του εμπορίου σε ό,τι αφορά τις σχετικές τάσεις, υψηλό πολύ είναι το έλλειμμα στο Μαλί. Οι εξαγωγές περιορίζονται σε λίγους μόνο εταίρους, εκτός από την ε, περιοχή της Δυτικής Αφρικής. Η Νότια Αφρική είναι, για παράδειγμα, ο μεγαλύτερος εταίρος της. Κάτι άλλο χαρακτηριστικό για τον εμπορικό κλάδο του Μαλή είναι ότι εστιάζεται σε δύο προϊόντα. Χρυσό καταρχάς 85% ε, και βαμβάκι. Αυτό έχει κάποιες συνέπειες. Αυτό φυσικά το υπογραμμίζουμε στην μελέτη, γιατί εξαρτάται πάρα πολύ από τα δύο αυτά αγαθά. Αυτό λοιπόν καθιστά τη χώρα πάρα πολύ ευάλωτη και ευαίσθητη σε διακυμάνσεις των τιμών. Και βλέπετε λοιπόν ότι μία από τις συστάσεις μας είναι διαφοροποίηση των εξαγωγών. Οι σε επενδύσεις πολύ καλά θα έχουν πάει και αυτό λοιπόν ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής. Η κυβέρνηση έχει εισαγάγει μία σειρά μεταρρυθμίσεων, κίνητρα που προσελκύουν τους μεγάλους επενδυτές οργανώσεις που και οργανώσεις που προωθούν τις επενδύσεις. Έχει σημειωθεί πρόοδος και στις υποδομές που είναι ασφαλώς πάρα πολύ σημαντικές για τις ε, επενδύσεις στο δικό δίκτυο, το ηλεκτρολιδωτικό δίκτυο έχει επεκταθεί και οι επενδυτές όμως εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, δυσκολίες ε, λόγω της ανεπάρκειας των υποδομών και ειδικότερα λόγω της υψηλής τιμής της ηλεκτροδότησης και των πόρων. Η γεωργία είναι εξαιρετικά σημαντική, είναι ένας από τους βασικότερους κλάδους της οικονομίας, 80% απασχολείται στο κλάδο αυτό του πληθυσμού. Ο κλάδος αυτός λοιπόν έχει τεράστιο δυναμικό επενδύσεων και σε ό,τι αφορά το βαμβάκι αλλά και σε ό,τι αφορά άλλα ε, προϊόντα, άλλα η παραγωγή των οποίων θα μπορούσε να επεκταθεί ή θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί για να αναπτυχθεί περαιτέρω ο κλάδος αυτός και σε άλλα τμήματα του πληθυσμού και ακόμα και σε περιόδους που αυξανόταν η παραγωγή του βαμβακιού αυτό είδαμε ότι δεν δημιούργησε νέες θέσεις απασχόλησης, δεν δημιούργησε νέες ευκαιρίες, κυρίως επειδή πρόκειται για προϊόν εξαγωγής. Όπως είπα αυτό ισχύει και για το χρυσό. Τονίζουμε λοιπόν το ότι η διαφοροποίηση έχει μείνει πίσω. Και ένας ε, από τους λόγους που έχει μείνει πίσω είναι το ότι η κυβέρνηση δεν έχει υποστηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επαρκώς. Αυτές λοιπόν δραστηριοποιούνται κυρίως στον άτυπο κλάδο και θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω η, κυβέρνηση. Τα ορυχεία επίσης είναι σημαντικά και η εξόρυξη χρυσού και εδώ βλέπουμε ότι τα πλεονεκτήματα δεν ε, ωφελούν όλο τον πληθυσμό, κυρίως επειδή η μεταποίηση και η επεξεργασία του χρυσού γίνεται στο εξωτερικό. Άρα και πάλι η μεγαλύτερη εξόριξη δεν οδήγησε σε δημιουργία θέσεων εργασίας και σε ανάπτυξη. Κοιτώντας ε, την, τον τομέα της απασχόλησης, τρία χαρακτηριστικά. Ε, χαμηλή δημιουργία θέσεων εργασίας, παρά την οικονομική ανάπτυξη, επέκταση του ανεπίσημου κλάδου εργασίας και αύξηση της ανεργίας κυρίως στους νέους. Αυτές οι τάσεις είναι ιδιαίτερα ανησυχητικέ. Προκαλούν κοινωνικές εντάσεις και αγανάκτηση στο κοινό. και οφείλονται σε έλλειψη πολιτικών για την ε, πάταξη αυτού του ανεπίσημου μαύρου κλάδου αν θέλετε, εργασία και την προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το Μαλί λοιπόν εξακολουθεί να είναι ένα από το, μία από τις πιο φτωχές ε, χώρες και στις διεθνείς κατατάξεις είναι στη θέση 182 από 187 χώρες σε ό,τι αφορά την τάση της φτώχειας. Φαίνεται ότι υπάρχει μία μείωση της φτώχειας, αλλά αυξάνονται τα νοικοκυριά και οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ε, πρόβλημα φτώχεια που ζουν κατά το όριο της φτώχειας. 5,7 εκατομμύρια το 2001, 6,4 το 2010. Ένα άλλο πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα είναι ανισότητες. Τεράστια προβλήματα, ιδιαίτερως ε, στις βόρειες περιοχές και σε ό,τι αφορά την, προ... πρόσβαση στην υγεία, την πρόσβαση στην παιδεία. Επίσης η επιστηστική κρίση το 2010 με την, στη μέση των τροφίμων ε, έπληξε ιδιαίτερα τις περιοχές αυτές. Κοιτώντας ε, τις δαπάνες στον κοινωνικό κλάδο, συνάδουν τα πράγματα με αυτά που παρατηρούμε και στις άλλες χώρες ε, της περιφέρειας κοιτώντας τις απάνες για την παιδεία. Βλέπουμε ότι αυτό αυξάνεται στα πιο εύπορα νοικοκυριά προγράμματα για τις χαμηλόμισθες κλίμακες είναι πολύ περιερισμένα. Φαίνεται λοιπόν ότι τα προγράμματα αυτά δεν φτάνουν στους, σε αυτούς που τα έχουν πιο πολύ ανάγκη από όλους δεν φτάνουν στους πιο φτωχούς, στα πιο φτωχά παιδιά, στα πιο φτωχά νοικοκυριά. Εντοπίσαμε μία σειρά ε, προκλήσεων σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Οι προκλήσεις αυτές έχουν επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης. Καταρχάς, ε, η έκθεση σε κρίσεις ε, σε διακύμανση των τιμών, επειδή βασικά, όπως σας είπα, επικεντρώνεται σε δύο προϊόντα τα οποία και εξάγει. Κοιτώντα τα τελευταία 7 χρόνια, η χώρα έχει αντιμετωπίσει τρεις ε, βασικές επιστικές ε, κρίσεις ε, και η διακυβέρνηση είναι χαμηλή από πλευράς της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά και την προσέλευση στις εκλογές μεγάλη διαφθορά. Το Μαλί στις διεθνείς κατατάξεις είναι από τις πιο διεφθαρμένες χώρες. Έχουν γίνει προσπάθειες να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή. Έχει δημιουργηθεί μια ειδική υπηρεσία η οποία εξετάζει περιπτώσεις διαφθοράς και τέλος η εγκληματική οικονομία, η οικονομία του εγκλήματος, ε, η αύξηση του λατρεμπορίου ναρκωτικών απαγωγών αποτελεί πλέον μια σημαντική πηγή εισοδήματος, ιδιαίτερα για ομάδες στο βόρειο τμήμα του Μαλή. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να το κατανοήσουμε πέρα από τη δυναμική της ε, απασχόλησης και της ανεργίας των νέων μάλλον σε συνάρτηση με την ενεργεία των νέων στην περιοχή εκείνη. Άρα οποιαδήποτε προσπάθεια να αντιμετωπίσει την οικονομική, τα οικονομικά θέματα του Μαλή θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ενεργείας. Γιατί σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν εναλλακτικέ ή πολύ περιορισμένε εναλλακτικέ πηγέ εισοδημάτων. Το Μαλί εξακολουθεί να είναι ένα από τα κράτη που χρειάζεται πιο πολύ ε, ανθρωπιστική βοήθεια στην υποσαχάρια Αφρική. Εξαρτάται από την ε, βοήθεια αυτή. Η ΙΠΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν τους μεγαλύτερους δωρητές, χορηγούς βοήθειας. Και τα βασικότερα ζητήματα είναι οι μεταφορές, η αποκέντρωση και πρόσφατα ξεκίνησε πιο έντονη συνεργασία με την Κίνα, την Ινδία και τη Λιβύη. Σε ό,τι αφορά τις ροές, θα γνωρίζετε ότι αναστάλησαν αυτές, ε, το μεγαλύτερο τμήμα της βοήθειας ανεστάλησε το 2012 μετά το ξέσπασμα της βίας και το πραξικόπημα της 22 Μαρτίου. Ωστόσο, ξαναξεκίνησαν μετά τη συμφωνία για τις ε, εκλογές του Ιουλίου του 2013 και η χώρα αναμένει σημαντική ροή βοήθειας τα επόμενα χρόνια. Το 2013 οι δωρητές ε, δεσμευτήκαν να χορηγήσουν πάνω από 3 δισεκατομμύρια ε, ευρώ για να υποστηρίξουν τα αναπτυξικά προγράμματα του Μαλή. Το Μαλή δραστηριοποιήθηκε πρόσφατα ιδιαίτερος σε περιφερειακές οργανώσεις, την Αφρικανική Ένωση, στην Οικονομική Ένωση των ε, ε, Δυτικοαφρικανικών χωρών. Συμμετέχει και στις σχετικές πρωτοβουλίες ε, των οργανώσεων αυτών για την παρακολούθηση της κατάστασης και μεταξύ άλλων παρακολούθηση των μακροοικονομικών όρων. Και επί της βάσης αυτής, για παράδειγμα το Μαλί, θεωρήθηκε μακροοικονομικά σταθερό, κοιτώντα τα ε, κριτήρια σύγκληση το Μάλι που ισχύουν στην περιφέρεια. Ε, το Μάλι συμμορφώνεται με τα πιο πολλά από αυτά τα κριτήρια. Το 2010 μόνο με δύο εξ αυτών δεν συμμορφώθηκε. Τέλος. Για το Μαλί αυτοί οι περιφερειακές σχέσεις είναι υψής της σημασίας λόγω της γεωγραφίας του, επειδή είναι περίκλειστη χώρα, αυτό σημαίνει ότι εξαρτάται ιδιαιτέρως από τους περιφερειακούς ε, διαδρόμους μεταφορών σε ό,τι αφορά την άντρεψη, σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, την υδρολεκτική ενέργεια. Χρειάζεται λοιπόν ε, συμφωνίες με τις γειτονικέ χώρες και αυτές οι σχέσεις θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω με τις όμορες χώρες ε, όπως τα ξέρετε από την κρίση και μετά σημειώθηκαν διάφορες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την οικονομία. Είναι σε ύφεση πλέον η οικονομία. Συρρυκνώθηκε η οικονομία λόγω της μείωσης των δωρεών που συνδείκνωσε διάφορους ε, οικονομικούς κλάδους και ασφαλώς επληκτική ο τουρισμός. και παρά την προστασία των κοινωνικών δαπανών στην υγεία και στην ε, παιδεία, όπου υποτίθεται ότι δεν έγιναν περικοπές, η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και της παιδείας έχει σοβαρά πληχθεί, ιδιαίτερο στο βορρά, όπου είναι ουσιαστικά υποδιάλυση. Και αυτό έχει μία σειρά επιπτώσεων. ιδιαίτερο ανησυχούμε για τα θέματα υγείας. Επίσης, περίπου 400.000 ε, εκτοπίστηκαν εσωτερικά. Μετακινήθηκαν, μετανάστευσαν προς τον Νότο. Για να κλείσω λοιπόν τώρα με, τα, με τις συστάσεις για την πολιτική. Για την οικονομία διαπιστώνουμε ότι παρά τις βελτιώσεις και αύξηση των κρατικών εσόδων, ε, πολλές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, και εκεί υπάρχει δυνατότητα για καλύτερη, πιο αποτελεσματική χρηματοδότηση των υποδομών και πιο αποτελεσματικές κοινωνικές πολιτικές ε, για επέκταση του κοινωνικού δικτύου. Και στη Γεωργία υπάρχει δυνατότητα για μεγαλύτερη διαφοροποίηση, κάτι που είναι θεμελιώδη σημασία για την οικονομία του Μάλι. Ε, να, γίνει ένα άνοιγμα της γεωργίας πέρα από το βαβάκι και σε άλλα τρόφιμα, ε, λαχανικά, φρούτα, ε, ελαιούχοι σπόροι. Έτσι θα αυξηθεί και η απασχόληση για να φανεί η γεωρική ανάπτυξη και η οικονομική ανάπτυξη και να φτάσει μέχρι τον κόσμο. Οι επενδύσεις θα συνεχιστούν, ήταν πολύ αποτελεσματικές στο παρελθόν στον τομέα εξόρυξη χρυσού. Σε ό,τι αφορά τι επενδύσει, κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει ή να ενισχυθεί στο μέλλον είναι η υποστήριξη τη κυβέρνηση προκειμένου να ανοίξουν κάποιες συμφωνίες για επαναδιαπραγμάτευση για έλεγχο, ώστε να συμπληρωθούν με απέτηση προς τους επενδυτές να κάνουν μελέτες κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κάτι που λείπει από τις υπάρχουσες συμφωνίες, θα μπορούσε να επανεισαχθεί μια τέτοια ρήτρα για να προωθηθούν επενδύσεις που θα είναι πιο ακριβοδίκες κοινωνικά και πιο βιώσιμες και περιβαλλοντικά. Επίσης θα πρέπει να δοθεί βοήθεια για να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι δωρητές ε, θα πρέπει να στηρίξει την κυβέρνηση στο να αντιμετωπίσει την ανεπίσημη οικονομία και να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες. Στη, στα ορυχεία, για παράδειγμα, μπορούν να προωθηθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για βιοτεχνική εξόρυξη και επιπλέον υπάρχει δυνατότητα για εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης ε, και για τους ανέργους. Ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αντιμετωπιστούν οι περιφερειακές ανισότητες. Τα πρόσφατα κυβερνητικά έγγραφα φαίνεται ότι υποβαθμίζουν ή παραβλέπουν αυτό το θέμα, αλλά όπως είπαμε οι βόρειες περιοχές του Μάλι βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση, έχει επιδεινωθεί το βιωτικό επίπεδο και μετά την κρίση υπάρχει σοβαρότατη ε, διάλυση, διακοπή διάλυση των κοινοφελών υπηρεσιών. Όλες αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να αποκατασταθούν ως κατά προτεραιότητα. Η διαφάνεια είναι επίσης σημαντικό στοιχείο γιατί έχω προγραμματιστεί τεράστια κονδύλια βοήθειας προς το Μαλί. Θα πρέπει να υπάρχουν αξιόπιστοι μηχανισμοί για να εξασφαλίσετε υποπτία της χρήσης των πόρων με συμμετοχή Κοινοβουλίου, μέσω μαζική ενημέρωση και κοινωνία των πολιτών. Επίση θα πρέπει να γίνει σωστή παρακολούθηση, αξιολόγηση και πρόθεση τη συγκέντρωση ε, δεδομένων, γιατί ελάχιστα γνωρίζουμε. Δεδομένα υπάρχουν μόνο για λίγου τομεί και ακόμα και εκεί που υπάρχουν δεδομένα η ποιότητά του είναι συζητήσιμη. Επίση θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την κυβέρνηση για να εφαρμόσει τη διαδικασία αποκέντρωση μέχρι στιγμής έχει εφαρμοστεί μόνο μερικώς. Και η τελευταία σύσταση πολιτικής ε, που περιλαμβάνει η μελέτη μας είναι μια ενθάρρυνση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει την περιφερειακή της προσέγγιση, κυρίως γιατί το Μαλί είναι περίκλειστη χώρα και υπάρχει δυνατότητα να ενισχυθεί η ανάπτυξη αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την κοινή διαχείριση των ε, πόρων της περιοχής. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο για την υιοθέτηση της περιφερειακής προσέγγισης. Θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή για να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι προκλήσεις και από τη χώρα την ίδια, αλλά και από την περιφέρεια γενικότερα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κάσμα πρώτα. Συγγνώμη, ο κύριος προηγείται. Α, συγγνώμη, ε, έχετε εσείς το λόγο. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ θερμά για την παρουσίαση της μελέτης. Ευχαριστώ και για τη μελέτη και για τις συστάσεις. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτησή μου αφορά τις δυνατότητες ε, για το fair trade, το δίκαιο εμπόριο. Το κύριο εξαγωγικό προϊόν είναι το βαμβάκι. Βέβαια υπάρχουν συστάσεις να γίνει διαφοροποίηση προς ε, οποροκυπευτικά και ελέγχους σπόρους. Θα μπορούσαν όλα αυτά τα προϊόντα να εμπίπτουν στο δίκαιο εμπόριο, στο fair trade. Υπάρχει λοιπόν περιθώριο εδώ για περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του τρόπου αύξηση ε, των εισοδημάτων των νοικοκυριών του Μαλή με το fair trade δηλαδή. Και η δεύτερη μου ερώτηση αφορά την κατάσταση στο Βορρά. Πολύ κακή διακυβέρνηση γίνεται στο Βορρά. Αυτό μπορεί να είναι, η κακή διακυβέρνηση μπορεί να είναι και αιτία αλλά και αποτέλεσμα της κρίσης. Επίσης, η πρόσβαση στις κοινοφελείς υπηρεσίες έχει επιδεινωθεί. Και είπαμε ότι η κατάσταση ε, στο Βορρά είναι χειρότερη, με αποτέλεσμα να ανθεί η οικονομία του εγκλήματος οι άνθρωποι παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και αυτενεργούν στη δικαιοσύνη. Βέβαια οι ενέργειες αυτές είναι παράνομες και κατά του κράτους, αλλά η κακή διαχείριση που ισχύει στο Βορρά, η κακή διακυβέρνηση, ίσως είναι όχι μόνο η ρίζα του κακού, αλλά και το αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής. Γιατί όσο χειρότερη είναι η διακυβέρνηση, τόσο μεγαλύτερη ένταση υπάρχει για αποκέντρωση, περισσότερες ένοπλες συγκρούσεις γίνεται. Πώς λοιπόν θα διαρρήξουμε αυτό το φαύλο κύκλο της ε, κακής διακυβέρνησης και της εγκληματικότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κατσμάρεκ. Euh, Μία ερώτηση όσον αφορά τους δείκτες σύγκλησης στη συγκεκριμένη ζώνη. Θα μας πείτε δύο λόγια για το θέμα. Είχα θέσει το ερώτημα και στην ε, Κομισιόν για τη Δυτική Αφρική. Πρόκειται για κριτήρια που συναρτώνται προς τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη και το δημοσιονομικό έλλειμμα, το έλλειμμα του προπολισμού. έχουν πετύχει πριν από στην περιοχή που ζηλεύουμε. Ο δείκτης όμως ανθρώπινης ανάπτυξης που βρίσκεται πέρα από τους ε, άλλους γενικούς οικονομικούς δείκτες. Ευχαριστώ. Κύριος Κατέσης Ελπίζω να το πρόφερα σωστά. Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ο κύριος Χατζησάβας, προφανώς. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν εκφράζω την ικανοποίησή μου για την έκθεση, διότι άπτεται των διευθυντικών προβλημάτων του Μαλή και δεν μιλάμε εδώ μόνο για το βόρα του Μαλή, έχουμε προβλήματα διακυβέρνηση που οδήγησαν στην γνωστή κρίση ζητήματα τα οποία πρέπει να πάρουμε υπόψη μας τα σοβαρά. Ο στόχος της αναβίωσης της χώρας είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και στις 15 Μαΐου του 2013 στη διάσκεψη των δωρητών που αναφέρθηκε άλλωστε προηγουμένω. Όπως υπογραμμίζετε και εσείς, η χώρα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εξωτερική βοήθεια εύκολα παρέχονται οι δημόσιες υπηρεσίες, βασίζεται η χώρα φυσικά στα ορυχεία και στον πρωτογενή τομέα, στην γεωργία κλπ. Πρέπει να δούμε λοιπόν αν μπορούμε να αναπτύξουμε επιπλέον νέους πόρους. Αυτό είναι στο τραπέζιο στο θέμα αυτή τη στιγμή. Δεύτερη γενική σκέψη. Η δημοσιονομική υπηρεσία, η ισορροπία με συγχωρείτε της χώρας. Ένα από τα βασικά μέσα που κινητοποίησαμε για να υποστηρίξουμε τις αρχές της χώρας να, να τη χώρα είναι ο δημοσιονομικός τομέας. Τι κάναμε. Ε, θα σας το περιγράψουμε δύο λόγια. Πρώτον, παρά την ένταση και την έκθεση της κρίσης που απειλεί το Μαλί, την ίδια του, την επιβίωση και το μέλλον του, παρά λοιπόν την σοβαρότερη της κρίσης που κατέστησε αναγκαία Ευρύτερη ξένη παρέμβαση, η κυβέρνηση δεν κατέρευσε ούτε το 2012 ούτε το 2013. Χάρη σε δύο λόγους. Πρώτον, η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών παρά τη διαφθορά στην οποία αναφερθήκατε είναι σχετικά καλή, ικανοποιητική στο Μαλί. Συμμερίζομαι τη γνώμη και άλλων διεθνών οργανισμών όπως το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, υπάρχει μια καλή ισορροπία, το χρέος δεν είναι υπερβολικό και η Άλλοι δείκτε δεν είναι κακοί όσον αφορά τη διαφάνεια, για παράδειγμα, τη διαδικασία κατάρτιση του προπολισμού και ούτω καθεξή. Όλα αυτά τηρούνται. Υπό αυτέ τι συνθήκε, το πλαίσιο λοιπόν τη δημοσιονομική διαχείριση, όπω είπα, είναι σχετικά ικανοποιητικό. Αυτό είναι και η εξήγηση. γιατί και πώ άντεξε το μαλλί. Δεύτερο λόγο, δεύτερη, δεύτερη εξήγηση, αν θέλετε, τη ε, αντοχής της χώρας και της κυβέρνησης είναι κάποιες καλές επιλογές που έγιναν κατά τη διάρκεια της ίδιας της κρίσης. Το 2012 συγκεκριμένα ο κρατικός προϋπολογισμός αναπροσαρμόστηκε χωρίς να ενσωματωθεί η ξένη βοήθεια στο σώμα του προϋπολογισμού. Δείγμα σύνεσης. Μειώθηκαν οι επενδύσεις, τα έξοδα λειτουργία στο δημόσιο σε πολύ μεγάλο βαθμό μάλιστα. Και έτσι άντεξε η κυβέρνηση πάνω από 18 μήνες παρά την σοβαρότητα, όπως είπα, της κατάστασης. Μετά από την επαναφορά της διεθνούς βοήθειας, ένας διορθωτικός προπολογισμός ε, ψηφίστηκε και περάσαμε σε μια πιο κανονική κατάσταση. Βάσει όλων αυτών λοιπόν λάβαμε την απόφαση να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε και το εργαλείο της δημοσιονομικής στήριξης. Τι κάναμε λοιπόν, εν προκειμένου. Λαβουμε φυσικά υπόψη μας τα, τους δείκτες, τα κριτήρια κλπ. Ε, τα οποία εννοείται θα εξετάσουμε στο πλαίσιο αυτό. Τι κάναμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, 220 εκατομμύρια ευρώ αλλά και 5 επιπλέον εκατομμύρια τεχνικής βοήθειας σε μακροπρόθεσμη βάση υπέρ του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και άλλων Υπουργείων του Μαλή που διαχειρίζονται αυτήν την εξωτερική βοήθεια. Τα κεφάλαια αυτά εκταμιεύθηκαν ήδη από την αρχή του 2013 μετά την διάσκεψη των δωρητών τον Μάιο του 2013. Τα κεφάλαια αυτά έδωσαν τη δυνατότητα στην κυβέρνηση της χώρας ενώπιση του 2014 να είναι πολύ πιο φιλόδοξη με στόχο ακριβώ να επαναδρομολογηθεί η ανάπτυξη και οι επενδύσεις. Επιπλέον, η τεχνική βοήθεια συνάδει πλήρω με τις νέες πολιτικές κατευθύνσεις, μεταξύ άλλων τον αγώνα κατά της διαφθοράς. Ελήφθησαν μέτρα, έγιναν έρευνες, τα ελεγκτικά όργανα έκαναν τη δουλειά τους, έτσι, η κυβέρνηση ικανοποίησε τις απαιτήσει των δωρητών όσον αφορά την διαφθορά, την μεταρρύθμιση της δημοσίας διοίκησης και το καθεξής. Μια κουβέντα μόνο για την διάσκεψη των δωρητών της 15 η Μαΐου. Δεν ήταν όλο μια πολιτική φιέστα, ξέρετε, ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Διότι κάναμε και άλλα πράγματα. Ακολούθησαν δύο υπουργικέ σύνοδοι. Την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες θα διεξαχθεί άλλη μια Υπουργική Σύνοδος και εκεί θα συζητήσουμε όλα τα κριτήρια επί των οποίων βασίζεται η βοήθεια που χορηγούμε. Οικονομικοί δείκτες, δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης κλπ. Θα συζητήσουμε τις υποδομές, τη συνολικότερη ανάπτυξη. Αυτά ακριβώς απαιτούμε και εμείς από την πλευρά μας στο νέο αναπτυξιακό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Μπαστάλη για να απαντήσει. Και να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις σας και τις προτάσεις, τα σχόλιά σας. Και τα σχόλια αυτά θα τα χρησιμοποιήσω στην αναθεώρηση και την διαμόρφωση της οριστικής μορφής έκθεσης. Σε ό,τι αφορά το fair trade, το δίκαιο εμπόριο ε, δεν αναφέρθηκε ίσως ε, ρητά, αλλά σίγουρα ισχύει αυτό. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό, ακόμη και στο τομέα του βαβακιού, αλλά και με την γεωργική διαφοροποίηση, με τη διεύρυνση σε άλλους γεωργικούς κλάδους, γιατί πραγματικά δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς το γεωργικό δυναμικό του Μαλή. <coughs> Βέβαια, το καλύτερο είναι να γίνει αξιοποίηση αυτή με δίκαιο και σωστό τρόπο και θεμητό. Σε ό,τι αφορά τα θέματα ε, αιτίου και αιτιατού, το αν η κακή διακυβέρνηση είναι η αιτία του κακού ή το αποτέλεσμα. Ισχύει αυτό που είπατε και η έξαρση της οικονομίας του εγκλήματος ε, οφείλεται στην έλλειψη ισχυρής παρουσίας της κεντρικής κυβέρνησης. Και η έξαρση αυτή όμως ενισχύει και την απουσία της κεντρικής κυβέρνησης. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει. Η πρόθεση αποκέντρωσης και η σχετική διαδικασία που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 90 στο τμήμα της διαδικασίας εκδημοκρατισμού σε μεγάλο βαθμό επέτυχε σημαντική πρόοδο. Δεν εφαρμόστηκε βέβαια στο έπακρο γιατί προσέκρουσε σε διάφορα προβλήματα και προκλήσεις η διαδικασία της αποκέντρωσης και ίσως ε, μερικές από τις τάσεις που επισημάναμε που ήταν και τα αίτια της ε, κρίσης, ίσως οφειλόταν στην ελληπή εφαρμογή της αποκέντρωσης. Όλοι πάντως αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στην ε, κλιμάκωση της βίας και της επακόλουθης πολιτικής κρίσης. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια σύγκλησης, η μελέτη περιγράφει τα κριτήρια σύγκλησης με στοιχεία για το Μαλί αλλά και στοιχεία για τις γειτονικές χώρες για να έχετε μια δυνατότητα να συγκρίνετε τις επιδόσεις του Μαλί σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Σε ό,τι αφορά το 2010, υπάρχει διαφορά στις επιδόσεις ανάλογα με τη χρονιά. Το 2010 το Μαλί υλοποίησε τα περισσότερα κριτήρια σύγκλησης. Το μόνο κριτήριο που δεν είναι η αναλογία εξωτερικού ισοζυγίου και ΑΕΠ και το λόγο προς τη φορολογία που είναι χαμηλότερος. Υπάρχει δυνατότητα και περιθώριο για το μαλλί να αυξήσει τη φορολογία του. Αρκετά ενδιαφέρον ε, συμπέρασμα αυτό. Πάντως μιλούμε για μακροοικονομικά κριτήρια σύγκλησης. Εξορισμού λοιπόν αυτή είναι η τομή στους οποίους γίνεται η παρακολούθηση παρακολούθηση και εποπτεία γίνεται και στο κοινωνικό τομέα, όχι στα πλαίσια αυτού του πλαισίου του οικονομικού, αλλά και περιφερειακά και διεθνώς έχουμε ειδικούς δείκτες για το Μαλί και οι βασικές τάσεις παρουσιάζονται στη μελέτη. Ευχαριστώ θερμά τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για τα σχόλιά του, πολύ ενδιαφέροντα σχόλια και θα τα λάβουμε υπόψη κατά την οριστικοποίηση της έκθεσης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Φραντσέσκα Μπαστάλη. Δόκτωρ Μπαστάλη. Η Ιταλίδα δεν είστε στο Βοκόνι σπουδάσατε. Αν μήπως θέλει κανείς το λόγο ε, να μας πει τίποτα ενδιαφέρον. Γιατί περιμένουμε τον Έλληνα Υπουργό και έχουμε χρόνο ελεύθερο. Αλλιώς μπορούμε να διακόψουμε προσωρινά ε, να πιούμε ένα καφέ, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να επιστρέψουμε για να μην δώσουμε κακή εντύπωση στον Έλληνα Υπουργό. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και περαιτέρω ερωτήσεις ε, στην κυρία Βαστάλη αλλά δεν βλέπω Άλλος κανεί θα θέλει το λόγο. Εσείς τι λέτε κύριε Γραμματεύ. Δεν έχετε γνώμη. Θέλει κανεί το λόγο. Ο γραμματέα μου λέει καλύτερα να διακόψω. Καλώ. Διακόπτουμε, θα πιούμε ένα καφεδάκι, αλλά δεν θα φύγουμε για να μην δώσουμε κακή εντύπωση στον Υπουργό. Πέντε παρα δέκα θα έρθει ο Έλληνας Υπουργός. Εμείς θα λίγο νωρίτερα για να τον περιμένουμε.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 Με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Κυριάκο Γεροντόπουλο, που είναι υφυπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων τη Ελλάδα, και θα μα παρουσιάσει τι προτεραιότητε τη Ελληνική Προεδρία ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα πλαίσια τη ανθρωπιστική βοήθεια. Πρώτα απ' όλα όμως ήθελα να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό τον κύριο Γεροντόπουλο για την καλοσύνη που είχε να έρθει στη συνεδρίασή μας και ελπίζουμε ότι και η δική σας Προεδρία όπως και οι προηγούμενες θα γίνει σε ένα πνεύμα στενής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στον τομέα των ανθρωπιστικών θεμάτων ε, θα έχουμε μια πληθώρα πολύ συγκεκριμένων προκλήσεων να αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες κρίσεις που είναι ιδιαίτερα σοβαρές, να εγκαινιάσουμε επίσης, να θεσπίσουμε το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας, ε, μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση των σχετικών διαπραγματεύσεων και να συνεχίσουμε και τις προσπάθειες για την αναθεώρηση του σχεδίου δράσεως του Χιόγκο για τη μείωση των ζημιών από θεομηνίες, να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να ενισχύσουμε τις καλές πρακτικές για θέματα ανθεκτικότητας κρίσης και να δούμε και το θέμα του συνδέσμου μεταξύ βραχυπρόθεσμης ανθρωπιστικής βοήθειας και μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής βοήθειας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Υφυπουργό για 20 λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, πολύ κύριε Πρόεδρε. Ειλικρινά είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν μου επιτρέπετε και μεγάλη συγκίνησή μου διότι ξανά είμαι εδώ πέρα στα έδρανα 25 χρόνια μετά. Για όσους δεν το ξέρουν, υπήρξε ένας από τους ευρωβουλευτές της πενταετίας 1984-1989 και τότε λέγανε ότι είμαι ο πιο μικρός ευρωβουλευτής ε, και πραγματικά εδώ σε αυτά τα έδρανα ε, για πέντε χρόνια έμαθα πολλά ε, συμπίωσα τις γνώσεις μου για την Ευρώπη και αγάπησα την Ευρώπη και πίστεψα πραγματικά ότι η Ευρώπη είναι το κοινό μας στο σπίτι. Βεβαίως στην εποχή εκείνη υπήρξαν κοντά, ήταν ευρωβουλευτές μεγάλα ονόματα δεν, θα, δεν θα ξεχάσω ποτέ τη Σιμών Βέιλ, η οποία είναι άλλωστε και η πρώτη πρόεδρος του εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ήταν συνάδελφος. Ε, ο Πιέρ Φλεμελέν, ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος του Κοινοβουλίου και μετά ο Λόρδος Πλάμπ, έτυχε να είμαι συνάδελφος με τον ε, Σπινέλη, το οποίο το όνομα φέρει αυτό το κτίριο. Έτυχε να είμαι ε, συνάδελφος με τον Βερλικουέρ, ο οποίος μετά από λίγους αποδίμησε και βεβαίω και τον Έλληνα τον Ευρυγένη, του οποίου η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμη και τώρα είναι σημείο αναφορά. Κοντά σε αυτού λοιπόν του ανθρώπου προσπάθησα και εγώ κάτι να μάθω και να είμαι σήμερα ξανά 25 χρόνια μετά εδώ. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να διαφωτίσω του συναδέλφου ε, ε, Ευρωβουλευτέ για τι θέσει τη Ελληνική Προεδρία επάνω στα θέματα τη ανθρωπιστικής βοήθεια, Μα πάνω απ' όλα θέλω να πω ότι Πιστεύω πραγματικά ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου του Ευρωπαϊκού είναι σημαντικός και οφείλουμε όλοι εμείς να κάνουμε τα πάντα για να τον ενισχύσουμε. Μόνο με ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ευρώπη θα προχωρήσει μπροστά. Και θα προχωρήσει μπροστά χωρίς τις παλινοδίες του παρελθόντος. Διότι χάθηκαν ευκαιρίες, οι οποίες ευκαιρίες σήμερα έχουν οδηγήσει ακριβώς σε αυτή την κρίση. Ε, λέω καμιά φορά ότι ως Ευρωβουλευτής, νέος Ευρωβουλευτής τότε, μετήχα στις διαδικασίες για το φόνο Τενεμπλό, για το φόνο Τενεμπλό και μετά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο υπήρξε συγητής τόσο της συνθήκης του Μάστριχ όσο και της συνθήκης της Λισαβόνος. Καμιά φορά χαριτολογώντας λέω ότι δεν υπήρξε εισηγητής της συνθήκης της Ρώμης γιατί τότε ήμουν αγέννητος. Αλλά παρόλα αυτά σας λέω ότι αυτή την Ευρώπη που είναι κοινό μας σπίτι οφείλουμε να την ενισχύσουμε όλοι μαζί και πάνω απ' όλα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ρόλο των Ευρωβουλευτών. Εδώ είναι η καρδιά της δημοκρατίας, επομένως ο Ευρωβουλευτής πρέπει να έχει περισσότερες αρμοδιότητες, να μπορεί να ελέγχει τα όργανα της κοινότητας και συγχρόνως ε, μεταφέροντας ακριβώς την πίστη, την πεποίθηση των, των, των πολιτών τους οποίους εκπροσωπεί, να μπορεί να δίνει δύναμη στην Ευρώπη, μια δύναμη η οποία σήμερα έχει χαθεί και ελπίζω στις ευρωεκλογέ που έρχονται να μπορέσουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις να ε, δώσουν το στίγμα τους και να πείσουν τους πολίτες ότι έχουμε ανάγκη από περισσότερη Ευρώπη, από περισσότερη ενότητα και έτσι μόνο θα μπορούμε να είμαστε ισότιμοι στα διεθνή φόρα, στι διαπραγματεύσει διαπραγματεύσεις οι οποίες γίνονται. Αυτά έτσι ως γενικές αρχές και μου επιτρέπετε να μπω κατευθείαν στο θέμα τώρα. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, Αξιότιμοι κυρίε συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, καταρχά θα ήθελα να εκφράσω την ευχαρίστησή μου για την ευκαιρία που μου δίνεται να παρουσιάσω σήμερα στην Επιτροπή ΝΤΕΒΕ τι προτεραιότητε τη Ελληνική Προεδρία στον ανθρωπιστικό τομέα κατά το τρέχον εξάμεινο. Η Ελληνική Προεδρία πιστεύει ακράδαντα ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεγάλων ανθρωπιστικών θεμάτων απαιτεί τη στενή συνεργασία του Συμβουλίου και της Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ε, αποτελεί άλλωστε και τον πλέον αντιπροσωπευτικό δημοκρατικό θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου από την Ελλάδα συμπίπτει με μια χρονική περίοδο για την οποία οι εκτιμήσεις είναι ότι οι ανθρωπιστικές ανάγκες σε τρίτες χώρες συνεπία φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών θα αυξάνονται ενώ οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι για την αντιμετώπιση τους συνεχώς μειούνται. Η ανάληψη ανθρωπιστικών δράσεων αποτελεί μία από τις πλέον απτές εκφράσεις των βασικών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και σε εποχή οικονομικής λιτότητας της, ε, της ευρωπαϊκής μας οικογένειας, που αποσχολεί ως γνωστόν έντονα και την Ελλάδα, η Ένωση εξακολουθεί να καθοδηγείται από τις αρχές του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της προσφοράς για την ανακούφιση των πλέον ευάλωτων πληθυσμών στην Ιφίλιο. Η Ελληνική Προεδρία είναι πεπισμένη ότι για εμάς τους Ευρωπαίους αυτό είναι ο καταλληλότερος τρόπος ανταπόκρισης στις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος τον 21ο αιώνα επακόλουθο το προαναφερθέντων είναι να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας αφού καλύπτει ετησίως το 50% περίπου της διεθνούς χρηματοδότησης για ανθρωπιστικούς λόγους. Για το 2014 η Επιτροπή έχει προϋπολογίσει να διαθέσει ποσό 874 εκατομμυρίων ευρώ ως ανθρωπιστική βοήθεια σε τρίτες χώρες συνεχίζοντας το σημαντικό έργο της Ιρλανδικής και Λιθουανικής Προεδρίας και έχοντας ταυτόχρονα ως γνώμονα την αρτιότερη προετοιμασία των εργασιών του επόμενου τρίου, ε, δηλαδή της Ιταλίας, της Λετωνίας και του Λουξεμβούργου, η Ελλάδα θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου η ανθρωπιστική βοήθεια της Ένωσης να παρέχεται έγκαιρα και αποτελεσματικά. Η ενίσχυση του συντονισμού προϋποθέτει ότι τα κράτη-μέλη θα προσπαθούν να καταλήγουν σε κοινέ εκτιμήσεις αναφορικά με τα δεδομένα και τις παραμέτρους μιας ανθρωπιστικής κρίσης, οι οποίες δίνονται να αποτυπώνονται και σε κείμενα κοινών μηνυμάτων που η ομάδα εργασίας Κοχάφα θα προωθεί στις αρμόδιες γεωγραφικές ομάδες του Συμβουλίου, την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας και στα κατά περίπτωση συναρμόδια όργανα της Ένωσης, ώστε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων να λαμβάνεται υπόψη και να συνεκτιμάται η ανθρωπιστική διάσταση με έναν πιο συστηματικό τρόπο. Η Ελληνική Προεδρία θα προωθήσει περαιτέρω την διασύνδεση και το στενό συντονισμό μεταξύ ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παρατηρούμενης μακρόφωνης ευπάθειας χωρών και πληθυσμιακών ομάδων που έχουν υποστεί φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Ο συνδυασμός ανακούφιση, αποκατάσταση και ανάπτυξη μέσω κατάλληλων μηχανισμών αφενός δημιουργεί συνθήκες διαρκούς ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων ή αστάθειας και αφετέρου εμπεδώνει κλίμα ομαλότητας και μετάβασης στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η μείωση της επικινδυνότητας των καταστροφών, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και η μετάβαση από τις ανθρωπιστικές κρίσεις στην ανάπτυξη αποτελούν βασικές προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας. Στο πλαίσιο αυτό θα θέσουμε ως ζήτημα έναρξη διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών της δυνατότητες προσφοράς του ιδιωτικού τομέα στην εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση ειδικών ανθρωπιστικών αναγκών, παραδείγματος χάρη διατροφικών, έχοντας ως προηγούμενο τα ήδη θετικά αποτελέσματα στον τομέα της ανάπτυξης. Ο ιδιωτικός τομέας είναι πιθανό να διαδραματίσει ένα πολύ χρήσιμο ρόλο στον εντοπισμό και την ένταξη νέων προϊόντων και διαδικασιών που ανταποκρίνονται σε εφιστάμενες λειτουργικές προκλήσεις και ευκαιρίες με στόχο την ταχύτερη ανάκαψη των πληγισών περιοχών καθώς και την μείωση της επικινδυνότητας των καταστροφών. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, Στη συνέχεια θα ήθελα να, να αναφερθώ πιο λεπτομερώς στις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας βάσει των παρακάτω τεσσάρων θεματικών ενωτήτων. Πρώτον, νομοθεσία, πρώτη ενότητα, νομοθεσία και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ανθρωπιστικό τομέα. Κανονισμός περί πρωτοβουλίας εθελοντών βοήθειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. European Union Aid Volunteers Initiative. Η Ελληνική Προεδρία θα ήθελε να ευχαριστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερος δε την εισηγήτρια κυρία Μισελ Στρίφλερ, την Επιτροπή, καθώς και τη Λιθουανική Προεδρία για το επικοδομητικό έργο τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με την οριστικοποίηση του κειμένου του σχεδίου κανονισμού για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας των εθελοντών βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή σας στις 17 Δεκεμβρίου του 2013. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως βάση την αποστολή εθελοντών κατόπιν προηγούμενης ε, προσεκτικής εκτίμησης των εκάστοτε επιτόπου αναγκών με στόχο η δράση τους να είναι ωφέλιμη τόσο για τους αποδέκτες της βοήθειας στο πεδίο όσο και για τους ίδιους τους εθελοντές. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Προεδρία προσβλέπει στην ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας με την υπερψήφιση του σχεδίου κανονισμού από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να ξεκινήσει η φάση υλοποίησης του. Επίσης, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, η Ελληνική Προεδρία πρόκειται να οργανώσει σχετικό συνέδριο στις Βρυξέλλες για να αξιολογηθούν οι ανάγκες των εκάστοτε εκτελεστικών εταίρων, δηλαδή των οργανώσεων αποστολής και υποδοχής εθελοντών. Β. Δεύτερον, ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ως γνωστόν, η European Consensus on Humanitarian Aid αποτελεί το θεμέλιο λίθο της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας της Ένωσης σε τρίτες χώρες στη βάση των αρχών του ανθρωπισμού, της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας. Η ελληνική Προεδρία θα παρακολουθήσει την αξιολόγηση της υλοποίησης του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής κοινή Αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια. Action Plan of the European Consensus on Humanitarian Aid κατά την περίοδο Ιουνίου 2008 Ιουνίου 2013. Στόχος είναι η μελλοντική βελτίωση του τρόπου εφαρμογής τόσο από την Ένωση όσο και από τα κράτη-μέλη. Η Ελληνική Προεδρία θεωρεί σημαντική την έκφραση των απόψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί των συμπερασμάτων και συστάσεων της εν λόγω αξιολόγησης. Σχέδιο δράσης για την ε, γάμα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της αθεκτικότητας σε χώρες επιρρεπείς σε ανθρωπιστικές κρίσεις. Η ελληνική προεδρία θα υποστηρίξει και θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγις την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ανθεκτικότητα που υιοθετήθηκε τον περασμένο Ιούνιο και καλύπτει την περίοδο 2013-2020. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πλέον ένα συγκεκριμένο στρατηγικό πλαίσιο μέσα από το οποίο θα μπορέσει να αναπτύξει αποτελεσματικές δράσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση διαδοχή της ανθρωπιστικής βοήθειας από αναπτυξιακά προγράμματα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο σε όλες εκείνες τις χώρες στις οποίες οι λαοί τους βιώνουν για χρόνια τις απάνθρωπες επιπτώσεις των παρατεταμένων ή επαναλαμβανομένων ανθρωπιστικών κρίσεων. Θα καταβάλουμε ιδιαίτερες προσπάθειες για την κατά το δυνατόν ουσιαστικότερη προώθηση του ενεξελίξη διαλόγου μεταξύ των αρμοδίων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Προς αυτή την κατεύθυνση και με γνώμονα την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης, η Ελληνική Προεδρία σχεδιάζει την πραγματοποίηση μιας άτυπης μικτής συνάντησης Κοχάφα, ΚΟΧΑΦΑ-ΚΟΝΤΕΒ... τον Ιούνιο του 2014 στην Αθήνα. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον και χρήσιμο να πληροφορηθούμε τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του σχεδίου αυτού. Πάμε στη δεύτερη ενότητα. Ανθρωπιστικές κρίσεις. Η ελληνική Προεδρία θα εργαστεί μεθοδικά ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξακολουθήσει να διαδραματίζει προεξάρχοντα ρόλο στην αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών ανθρωπιστικών κρίσεων παγκοσμίω, ιεραρχώντας ως άμεση προτεραιότητα, βάσει των σημερινών δεδομένων, την Συρία και τις γειτονικές της χώρες, την Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία και τον Νότιο Σουδάν. Παράλληλα, θα μεριμνήσουμε να διατηρηθεί η δυναμική ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παρατεταμένες και ξεχασμένες κρίσεις. Π.χ. Αφγανιστάν, Μιαμάρ, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Κολομβία, Κέρας της Αφρικής, περιοχή Σαχέλ κλπ. Οι οποίες συχνά επισκιάζονται από την ξαφνική εμφάνιση κρίσεων όπως ο τυφώνας που έκλειξε τις Φιλιππίνες τον περασμένο Νοέμβριο με την περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής θα επιδιώξουμε να ενισχύσουμε την υπεράσπιση της αναγκαιότητας των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων έναντι κυβερνήσεων τρίτων χωρών προκειμένου να συμβάλλουμε στη δημιουργία των συνθηκών για μια αποτελεσματική και αποδοτική παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς όφελος των εκάστοτε πλητωμένων. Θα ήθελα επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική προεδρία θα παραμείνει σε στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή καθώς και τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών όπως ΟΤΣΑ, ΔΕΕΦΠ, ε, UNICEF καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων σε σχέση τόσο με τις επίγουσες όσο και τις παρατηταμένες ανθρωπιστικές κρίσεις ανά την Ιφίλιο. Τρίτη ενότητα, είναι οι πρακτικές και λειτουργικές προκλήσεις στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Όσον αφορά στη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, η ελληνική Προεδρία θα ενισχύσει το στρατηγικό συντονισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεγιστοποιώντας έτσι την αποτελεσματικότητά της. Τούτο απαιτεί τον εντοπισμό τυχών κενών, την αποφυγή ενδεχομένων επικαλύψεων, καθώς και την καλύτερη διασύνδεση της ανθρωπιστικής με την αναπτυξιακή και την μακροοικονομική χρηματοδοτική βοήθεια. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεχίσουμε την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις πλέον πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας της Ένωσης. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η πρόσβαση της βοήθειας σε όσους την έχουν ανάγκη, η ασφάλεια του ιατρικού προσωπικού και των μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων, καθώς και ο σεβασμός των αρχών του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Η Ελληνική Προεδρία χαιρετίζει τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σημερινές προκλήσεις στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας και προσβλέπει σε μελλοντικές ανταλλαγές απόψεων επ' αυτού του θέματος. Η Ελληνική Προεδρία θα παράσχει το απαιτούμενο πλαίσιο για το συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να διασφαλίσει ότι οι απόψεις της ως κύριου χορηγού ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίω θα συμπεριλαμβάνονται στις διάφορες ανεξελίξει διεθνείς πρωτοβουλίες και αναφέρονται δικτικά. Το πλαίσιο δράσης μετά το Χιόγκο που αποβλέπει στη συνεχή βελτίωση των εθνικών και διεθνών μηχανισμών αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών καθώ και στη μείωση τη επικινδυνότητάς του, Την ομάδα στήριξη δωρητών του ΟΤΣΑ τη μεταρρυθμιστική ατζέντα για την ενίσχυση του διεθνούς ανθρωπιστικού συστήματος από πλευράς των ΗΕ. Η ελληνική Προεδρία θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις προετοιμασίες για τη σύγκληση της πρώτης παγκόσμιας ανθρωπιστικής συνόδου κορυφής το 2016. Αν και είναι πολύ νωρίς για την επεξεργασία συγκεκριμένων κοινών θέσεων της Ένωσης για τη Σύνοδο Κορυφής, εντούτοις θα βοηθήσουμε στη διευκόλυνση του συντονισμού στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκής ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για να αποτελέσει βασικό παράγοντα στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της Συνόδου Κορυφής. Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας, θα ήθελα να επαναλάβω ότι προβλέπουμε και αναγνωρίζουμε τη σημασία του διαλόγου μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξέβρεση του καλύτερου δυνατού τρόπου διαμόρφωσης ενός αποτελεσματικού διεθνούς ανθρωπιστικού συστήματος στα χρόνια και τις δεκαετίες που έρχονται. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Ευχαριστώ. κύριε Υπουργέ. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Γκέρενς ε, θα ήθελε το λόγο. Κύριε Γκέρενς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε αμέσως το λόγο, γιατί δυστυχώς ε, θα θέσω την ερώτηση, θα περιμένω την απάντηση και αμέσως μετά θα φύγω, γιατί έχω μια ανηλυμένη υποχρέωση στο Λουξεμβούργο στις 8 η ώρα σήμερα το βράδυ. Ακούσαμε τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας, έχω διάφορα σχόλια. Καταρχήν να χαιρετίζω τον επικοδομητικό τόνο της εισαγωγικής σας ομιλίας στην Επιτροπή Ανάπτυξης, κύριε Υπουργέ. Εν συνεχεία, θα ήθελα να πω ότι από την αρχή της κοινοβουλευτικής θητείας έχουμε διανύσει αρκετό δρόμο. Στην αρχή δεν είχαμε σχεδόν καμία επαφή με την χώρα που ασκούσε την Προεδρία του Συμβουλίου. Σε ό,τι αφορά με τις επαφές με τον αρμόδιο Υπουργό για θέματα συνεργασίας. Και η Ελληνική Προεδρία συμπίπτει με μια δύσκολη κοινοβουλευτική περίοδο γιατί έχουμε ακόμη δύο-τρεις συνδιαλλαγές που δεν είναι ιδιαίτερα επίμαχες. Δεν έχουμε τίποτα φλέγων και γι' αυτό μπορούμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στις πολιτικές πτυχές για τους λίγους μήνες που μας έχουν απομείνει μέχρι τις ευρωεκλογέ. Χθες είχαμε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων με τον αρμόδιο της ε, ε, ανθρωπιστικής δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μας μετέφερε τις δυσκολίες χρηματοδότησης, όπως μας εξήγησε και η αρμόδια Επίτροπος. Μας διαβεβαίωσε όμως ότι θα είναι ε, παροδικές αυτές οι δυσκολίες χρηματοδότησης. Όταν έχουμε επαρκή δημοσιονομικά μέσα, μπορούμε να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις χρηματοδότησης. Είχα προτείνει χθε στην ε, Επιτροπή να στραφεί προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να ζητήσει μία προχρηματοδότηση για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες ρευστότητας που ενδεχομένως αντιμετώπιζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση των ανθρωπιστικών δράσεων. Μια και όμως ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, ε, συνδέεται με τα κράτη-μέλη, με τα κράτη-μέλη, θα ήθελα να συστήσω στην Ελληνική Προεδρία να εξετάσει αυτό το θέμα και να δούμε σε ποιο βαθμό θα μπορούσαμε να υπερβούμε τις παροδικές αυτές δυσκολίες ρευστότητες που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απευθυνόμενη προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ούτε στο Κοινοβούλιο, ούτε στη δική μας Επιτροπή κανένας δεν θα ήταν κατά μιας τέτοιας ε, ενέργειας για να ξεπεράσουμε τη δυσκολία αυτή. Επίσης ε, γνωρίζω ότι έχετε στενές σχέσεις και με τις επόμενες προεδρίες που είναι ένας πολύ καλής τρόπος για να εξασφαλιστεί μια συνέχεια των δράσεων σε ό,τι αφορά την ε, συνεργασία και την ανάπτυξη και χαίρομαι για την ε, ανταλλαγή απόψεων που έχουμε με την Ελληνική Προεδρία, γιατί στο παρελθόν τέτοιου είδου διάλογο ήταν αδύνατο. Ευτυχώ έχουμε αφήσει πίσω μα αυτή την περίοδο έλλειψη επικοινωνία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Κατσμάρεκ. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ τον ε, κύριο Υπουργό για την προθυμία του, για την συνάντηση που είχαμε και για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας και για τα πολύ καλά και ευγενικά του λόγια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ δύσκολο να μιλούμε για προτεραιότητε σε αυτή την φάση τη θητεία, γιατί όταν μιλούμε για επιχειρησιακέ ε, δράσει, ε, δεν ε, μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων πού θα εμφανιστούν οι ανθρωπιστικέ ανάγκε. Υπάρχουν όμω μερικέ συγκρούσει και μερικέ κρίσει που γνωρίζουμε ήδη. Συρία, Νότιο Σουδάν, για παράδειγμα κεντροαφρικανική δημοκρατία και γνωρίζουμε ήδη ότι υπάρχουν ανθρωπιστικές ανάγκες. Έχω δύο ερωτήσεις. Μας μιλήσατε για την ασφάλεια του προσωπικού στον ανθρωπιστικό τομέα. Τέτοια προβλήματα έχουμε κάθε χρόνο και αυτή τη στιγμή στο Νότιο Σουδάν πολύ συχνά τα προβλήματα δεν είναι ούτε οικονομικά ούτε βοήθειας το θέμα είναι ότι εξαιτία τη έλλειψη ασφάλεια δεν, δεν μπορεί να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια σε μερικέ ζώνε που χυμάζονται από τέτοια ένοπλη σύγκρουση. Και μερικέ φορέ έχουμε και απώλεια ζώων του ανθρωπιστικού προσωπικού. Τι σκέφτεται να κάνει η ελληνική προεδρία ώστε να ενισχύσει αυτή την ασφάλεια για το προσωπικό της παροχής της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά τις ανθρωπιστικές ανάγκες ε, και τις χώρες που πρέπει να τις εξαναγκάσουμε ουσιαστικά για να δεχτούν την ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί υπάρχουν ε, χώρες που είναι ε, απρόθυμες να δεχτούν ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ έχουν ανθρωπιστικές ανάγκες. Για παράδειγμα η Βόρεια Κορέα. Γίνονται κάποιες απόπειρες να βοηθήσουμε τέτοιου χώρες που είναι όμως κλειστές και απρόθυμες. Πώς μπορούμε να παροτρύνουμε αυτές τις χώρες για να κάνουν ένα άνοιγμα για μεγαλύτερη συνεργασία. Ευχαριστώ. Grazie. L'onorevole Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εσάς ε, κύριε πρόεδρε από τη Συμβουλίου που ήρθατε εδώ πέρα σήμερα να μας παρουσιάσετε τα σχέδιά σας για το επόμενο εξάμεινο, γιατί πράγματι αυτό έχει καταστεί πλέον ε, έθιμο και πιστεύω ότι είναι και σημαντικό και σωστό. Την τελευταία εβδομάδα ο κυβερνών κ. Σαμαράς ήρθε στη, στο Στρασβούργο και μας παρουσίασε την κατάσταση στην Ελλάδα και ξεκαθάρισε στους ευρωβουλευτές ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει πλέον η Ελλάδα και ότι αναγνωρίζεται σε μεγάλο βαθμό το Κοινοβούλιο και ότι λαμβάνονται από κοινού οι αποφάσεις με το Κοινοβούλιο. Είναι καλό το γεγονός ότι στην Προεδρία σας επικεντρωνόσαστε στην ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί όντως τα τελευταία χρόνια έχει ανακύψει ως ένα πολύ σημαντικό σημείο για το οποίο διατίθονται περιορισμένοι πόροι συνολικά. Εν ώψη της κρίσης της Συρίας, στο Νότιο Σουδάν, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στο Μαλί, θα πρέπει να προσθέσω, μιας και συζητήσαμε πριν από λίγο για το Μαλί. Εν ώψη λοιπόν των κρίσεων αυτών, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε σε τέτοια ζητήματα. Θα μου άρεσε ιδιαίτερα η ιδέα ενός βοηθητικού μηχανισμού για τα κράτη-μέλη. Να προσταθεί λοιπόν και αυτό ως ιδέα στην συζήτηση. Η Επιτροπός Γεωργίευα κάθε φορά που ανακύπτει μια κρίση ή που οξύνεται μια κρίση, ουσιαστικά περνάει και ζητιανεύει από τα κράτη-μέλη και ζητού, ζητάει χρήματα. Μία λοιπόν πρόταση ήταν η Ευρωπαϊκή απο τα κρατη μελη και ζηταει χρηματα Τράπεζα αλλά πιστεύω ότι αν υπήρχε ένας ε, τέτοιος μηχανισμός ε, βοηθητικός που θα ε, επιβάρυνε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με την οικονομική τους ισχύ, θα ήταν τα πράγματα πιο απλά. Το κάνουμε αυτό για τη διάσωση των τραπεζών. Γιατί όχι και σε θέματα αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων. Μιλήσατε για το θέμα το νομοθετικό. Χαίρομαι που μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντών και πιστεύω ότι από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε, ε, έχουμε θέση στα πόδια της, έχουμε δημιουργήσει αυτή την υπηρεσία εθελοντών και θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο. Γιατί ολοκληρώνεται τη θητεία της ε, η τρέχουσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άρα θα ήταν πάρα πολύ ευπρόσδεκτο μέχρι τότε να έχει ολοκληρωθεί και το σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντών. Με την ανθρωπιστική κρίση και λόγω της εγκύτητας με τη Συρία έχουμε προσεγγίσει το θέμα. Μιλήσατε για το θέμα της μετανάστευσης που περνάει και μέσα από την Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο μέσα από την Ιταλία, από την Λαμπεντούζα. Μιλήσατε για την ευθύνη της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης για τη Συρία. Τελευταίο σημείο κριτικής το οποίο θέλω να θίξω. Οι αιτήσιες συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα 78 κράτη της ε, ΑΚΕ. Η εκάστοτε Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, φιλοξενεί και την σύνοδο με τις χώρες ΑΚΕ. Αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Η Ιρλανδία όμως ήταν η πρώτη χώρα που αρνήθηκε να διεξαγάγει για οικονομικούς λόγους την ε, συνέλευση αυτή στην Ιρλανδία. Η ελληνική κατάσταση, η κατάσταση της Ελλάδας είναι ακόμα πιο δύσκολη από ότι ε, αυτή της Ιρλανδίας, αλλά θα το καλωσόριζα εάν δείχνατε αλληλεγγύη προς τις 78 αυτές χώρες ΑΚΕ και διοργανώνατε την συνέλευση αυτή στην Ελλάδα. Τα πιο πολλά χρήματα, οι πιο πολλοί πόροι διατίθενται από ευρωπαϊκής πλευράς άλλωστε και νομίζω ότι θα ήταν μια άσχημη ένδειξη προς τις χώρες ΑΚΕ αν εμείς ε, από πλευράς Ευρώπης, αν η εκάστοτε Προεδρία δεν κατάφερνε να διοργανώσει αυτή την ε, συνέλευση στην οποία συμμετέχουν ε, βουλευτές από πάνω από 100 χώρες. Αυτό για να αποφευχθεί ενδεχομένως τη μελλοντική προεδρία, δεν ξέρω σε ποια χώρα θα είναι η προεδρία σε, μια, σε ένα έτος, για να αποφύγουμε την κατάσταση κατά την οποία θα αρνηθεί και η επόμενη προεδρία. Χώρες όπως η Αιθιοπία, ε, το Τογκό, όταν τέτοιες χώρες με πόνο καρδιάς και με το αίμα τους πληρώνουν για να διοργανώσουν τέτοια συνέλευση, νομίζω ότι θα ήταν τουλάχιστον καθήκον μας και εμείς από την πλευρά Ευρώπη Ευρώπης να διοργανώσουμε κάτι αντίστοιχο. Μάλιστα, θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Υπουργό για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ε, η Ελληνική Προεδρία ευθύς εξ αρχής έχει θέσει σαν βασικό της στόχο την συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πραγματικά εμείς είμαστε μια χώρα η οποία πιστεύει στην ε, ενοποίηση της Ευρώπης. Είμαστε από εκείνες τις χώρες, η δέκατη που μπήκα μέσα στην, ε, ε, στην τότε ΕΟ και σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση, που από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε όμως δώσαμε αγώνα για την εμβάθυνση των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι περισσότερες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόσο ε, στο τομέα της, της δυνατότητας παραγωγής νομοθετικού έργου όσο και στον ελεκτικό ε, για την Ευρώπη θα είναι ε, μια, ένα κέρδος διότι έτσι οι λαοί της Ευρώπης, οι πολίτες της Ευρώπης θα έχουν δυνατότητα να εκφράζονται μέσω του Κοινοβουλίου, να λένε τη φωνή τους και τις απόψεις τους. Επομένω είναι ξεκάθαρο ότι εμεί θέλουμε να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό θα κάνουμε. Στη συνέχεια θέλω να σα πω ότι αυτή η διαδικασία που λέτε, τουλάχιστον επί δικών μου ημερών δεν υπήρχε. Η Προεδρία δεν έρχονταν ούτε στι επιτροπέ ούτε στην Ολομέλεια. Ε, βεβαίως, όπως λένε κάποιοι συνεργάτε μου, εγώ είμαι, ήμουν Ευρωβουλευτή τον προηγούμενο αιώνα και ίσω οι απόψει τότε είναι, ε, ήταν τελείω διαφορετικέ από αυτέ που είναι σήμερα αλλά και πάλι θεωρώ ότι τα βήματα τα οποία έχουν γίνει με τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι βήματα μικρά. Και επειδή είμαι γιατρός, καμιά φορά χρησιμοποιώ και κάποιους όρους βιολογίας, ιατρικής, ήταν μια, την, χαρακτηρίζω ως οπισθόδρομο εξέλιξη. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάει πιο μπροστά, χάσαμε την ευκαιρία, επομένως αυτό είναι κάτι το οποίο το βρίσκουμε μπροστά μας με τις διάφορες κρίσεις οι οποίες δημιουργούνται. Ε, θέλω λοιπόν τώρα να μπω στις ερωτήσεις σας οι οποίες πραγματικά είναι εξαιρετικές. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να σας ικανοποιήσω για όλα αυτά. Δεν, πρέπει να σας πω ότι με το θέμα της των ε, ανθρωπιστικών κρίσεων είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι. Έχω εξαιρετικούς συνεργάτες οι οποίοι με βοηθούν, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι απόλυτος γνώστης αυτών των θεμάτων. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω να σας απαντήσω και συνάδελφοι από το Λουσέβου, θέλω να σας πω ότι πραγματικά ε, σχετικά με τις, ε, αναφορικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών των ανθρωπιστικών εταίρων από πλευράς της Γενικής Διευθύνσεως της ΕΚΟ και το ενδεχόμενο ανάγκης αυξήσεως του επίπεδου πιστώσεων πληρωμών της ΕΚΟ, η Ελληνική Προεδρία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, παράσχει στο Συμβούλιο, να δώσει στο Συμβούλιο την απαραίτητη ενημέρωση και αυτό θα γίνει στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Κοχάφα 23 και 24 ε, Ιανουαρίου. Η Προεδρία πρόκειται να ενημερωθεί λεπτομερώς από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Σόρενσεν, για την προβλεπόμενη πορεία εκτέλεσης του προπολογισμού του 2014 και το ενδεχόμενο να επηρεαστεί αρνητικά η υλοποίηση ανθρωπιστικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γενική Προεδρία πρόκειται να εξετάσει από κοινού με τα κράτη-μέλη τρόπους συστηματικής παρακολούθησης του εν λόγω ζητήματος. Ε, ως το θέμα της προάσπισης βασικών ανθρωπιστικών αρχών και αντιμετώπιση προκλήσεων πρόσβαση ανθρωπιστική βοήθεια και ασφάλεια προσωπικού. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, κύριε συνάδελφε, αυτό. Πραγματικά βλέπουμε καθημερινά εκπροσώπου φορέων που πηγαίνουν στι χώρε για να παράσχουν βοήθεια να πάγονται, να δολοφονούνται, να κινδυνεύουν σίγουρα. Η Ελληνική Προεδρία υποστηρίζει πλήρω τι αρχέ ανθρωπισμού, ανεξαρτησία, αμεροληψία και ιδιωτερότητα τη ανθρωπιστική βοήθεια. Πρόσφατε ανθρωπιστικέ κρίσει στην ΑΕΤ το 2010, στι Φιλιππίνες το 2013, στη Συρία, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στο Σουδάν, αναδεικνύουν μέγεθο και εύρο ανθρωπιστικών προκλήσεων, τι οποίε καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σήμερα, καθώ και αυξανόμενη δυσκολία προάσπιση βασικών ανθρωπιστικών αρχών, πρόσβασης ανθρωπιστικής βοήθειας και διασφάλισης προστασίας προσωπικού ανθρωπιστικών επιχειρήσεων. Η Ελληνική Προεδρία, η Ελληνική Προεδρία θα συνεχίσει προσπάθειες προηγουμένων Προεδριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσουν την προάσπιση των βασικών ανθρωπιστικών αρχών και να διασφαλίσουν την προστασία του προσωπικού των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων. Για μένα είναι βασικό αυτό εδώ. Εάν δεν διασφαλίσουμε την προστασία του προσωπικού, τότε είναι αδύνατον να πετύχουμε τους στόχου μας με την ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αρχή δεν θα μπορεί να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια και στα επόμενα στάδια δεν θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν να πάνε και να βοηθήσουν. Κρίνουμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί πρώτον με τη χρήση και, με τη χρήση και τη συμπληρωματικότητα του συνόλου των εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση κρίσεων επί εδάφους τρίτων χωρών. Δεύτερον, με την ενίσχυση συνεργειών σε επίπεδο προγραμματισμού και διάθεσης πόρων και τρίτον, με την ενίσχυση του συντονισμού ανθρωπιστικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντίστοιχες δράσεις των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών ανθρωπιστικών οργανισμών και υπηρεσιών. Όπως ξέρουμε, ο ΙΕ έχει πολύ μεγαλύτερο δίκτυο από ό,τι έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλο τον κόσμο. Επομένω, πολλέ φορέ η ανθρωπιστική βοήθεια την οποία στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνεται, φτάνει στον προορισμό τη μέσω καναλιών του, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που άλλωστε και τα, ε, όλα τα μέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και μέλη του, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και η συνεργασία σε, αυτό το τομέα του, ε, τουλάχιστον είναι απόλυτη και σίγουρη. Ταυτόχρονα, η Ελληνική Προεδρία θα επιδιώξει να συζητήσει διεξοδικά, συστηματικά και με στρατηγικό προσανατολισμό με το σύνολο των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύο βασικά θέματα. Πρώτον, τη βελτίωση παροχής διασυνοριακής, αυτό cross-border, και ανάμεσα σε εμπόλεμες ζώνες, το cross-line ανθρωπιστικής βοήθειας και δεύτερον, απρόσκοπτη πρόσβαση και προστασία του ανθρωπιστικού χώρου. Στόχος της ελληνικής προεδρίας για τα ανωτέρα θέματα θα είναι η επεξεργασία σχετικών κατευθυντήριων γραμμών τα οποία θα εγκριθούν από το Συμβούλιο κατά προτίμηση έως τέλος του Ιουνίου του τρέχοντος έτους, δηλαδή επί, ελληνικής, ε, επί του εξαμήνου της ελληνικής προεδρίας πώς η ελληνική προεδρία σκέφτεται να, να ανταποκριθεί στις πιο πάνω ε, προκλήσεις. Καταρχάς πρωτοκαθεδρία και προβάδισμα σε σχεδιασμό και διάθεση ανθρωπιστικών κονδυλίων η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, όπως βεβαίως γνωρίζετε, ε, μάλλον την πρωτοκαθεδρία και το προβάδισμα στο σχεδιασμό και στη διάθεση ανθρωπιστικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει, όπως όλοι γνωρίζουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ρόλος της εκάστοτε Εθνικής Προεδρίας είναι να συνδράμει επικοδομητικά σε αυτές τις προσπάθειες και σε αυτές τις ανθρωπιστικές δράσεις της Επιτροπής. Η Ελληνική Προεδρία γνωρίζει επίσης ότι η καλή συνεργασία ε, του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο επιτυχίας της ανθρωπιστικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να επιτύχουμε απτά, συγκεκριμένα και άμεσα αποτελέσματα και να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις στις πιο πάνω προκλήσεις. Το πλαίσιο αυτό αποτελεί βασική μέρημνα της ελληνικής προεδρίας και επομένως στόχος μας είναι ο σχεδιασμός του προγραμματισμού ανθρωπιστικών δράσεων που να προάγει συνέργειες και αλληλοσυμπήρωση κοινών δράσεων και επίσης ο συντονισμός με διεθνείς παρόχους ανθρωπιστικής βοήθειας είπα κάτι προηγουμένως, περιοχή. Η ελληνική, η ελληνική Προεδρία αναμένει με ενδιαφέρον τι προτάσει του Ευρωκοινοβουλίου, τι προτάσει όλων μα για το πώ μπορούν να ξεπεραστούν οι πιο πάνω προκλήσει και προτίθεται, όπω το έχω πει και προηγουμένω και θα, θα το λέω συνεχώ να συνεργαστεί η Ελληνική Προεδρία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προ την υλοποίηση του στόχου αυτού. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τίποτε δεν μπορεί να προχωρήσει στην Ευρώπη χωρίς τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό αποτελεί την καρδιά του, ε, αυτής της Ένωσης και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Ο προπολογισμό τώρα τη ανθρωπική βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω ξέρετε, σύμφωνα με το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, ο προπολογισμό τη ανθρωπιστική βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο των 7 επομένων ετών, αρχή γενομένη από την Ελληνική Προεδρία, ανέρχεται σε περίπου 5,9 δισεκατομμύρια σε τιμές του 2011. Περίπου δηλαδή 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε σύγκριση με το προηγούμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο του 2007-2013 έχουμε μια αύξηση της τάξης του 2,8%. Σε μια περίοδο παρέτηταμένη δημοσιονομικής δυσχέρειας, η διατήρηση του προπολογισμού σε επίπεδα ανάλογα με την προηγούμενη δημοσιονομική περίοδο αποτελεί μια σαφή ένδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί υψηλά στην ατζέντα της την παροχή αλληλεγγύης σε πληθυσμού που έχουν ανάγκη διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Ως εκ τούτου, επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιθανό να παραμείνει ο σημαντικότερος χορηγό στον κόσμο παρέχοντας περίπου το 50% της παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας. Στοχεύουμε βεβαίως και στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και ποιότητας της ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της βελτίωσης του συντονισμού και της αποφυγής αλληλεπικαλύψεων ανθρωπιστικών δράσεων της ε- ε- ε- Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπολείπων οργάνων. Εγώ από, από εκεί και πέρα θέλω να σας πω και κάτι εγώ, Επειδή τέθηκε ένα σημαντικό ζήτημα για την ε, εάν θα γίνει ή όχι η συνεδρίαση της ε, κοινή κοινωνικής συνέλευσης Αφρικής Καραϊβικής Ελληνικού και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα ή όχι, θα σας πω το εξής. Είναι γεγονός ότι για πολλά χρόνια αποτελούσε πρακτική. Από το, αν θυμάμαι καλά, από το 2003. Ε, αν θέλετε, παράδοση είναι αποτελούσε ε, πρακτική να γίνεται συνεδρία τη κοινή κοινοβουλευτική ε, συνέλευση Αφρική, Καραϊβική και Ελληνικού... και Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο εξάμεινο στη χώρα που ασκούσε την προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρακτική αυτή διακόπηκε πέρσι από την Ιρλανδία. Η ελληνική προεδρία έχει σαφή άποψη και βαθιά εκτίμηση για το έργο και τη σημασία τη συνέλευση. Για το λόγο αυτό προσπάθησε να διατηρήσει την πρακτική αυτή. Δυστυχώς όμως δημοσιονομικοί και οργανωτικοί περιορισμοί κατέστησαν την επιθυμία αυτή να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική προεδρία δεν θα ανταποκριθεί και δεν θα παράσχει στη συνέλευση κάθε δυνατή βοήθεια. Σας διαβεβαιώ ότι θα το πράξει αποδίδοντας τον οφειλόμενο σεβασμό γιατί θεωρούμε ότι η δουλειά την οποία κάνει η συνέλευση είναι σημαντική. Το ότι δεν θα γίνει στην Αθήνα ή εντό του ελληνικού χώρου δεν σημαίνει ότι θα χάσει την αξία τη και τη σημαντικότητά τη. Άλλωστε και στι Βρυξέλλε που έγινε πέρσι επί Ιρλανδική Προεδρία τα αποτελέσματα ήταν θετικά και νομίζω ότι και οι εκπρόσωποι των χωρών τη Αφρική, τη Καραβική και του ελληνικού έμειναν ικανοποιημένοι όχι για, για τον τόπο, οι Βρυξέλλε είναι υπέροχη πόλη, ε, όχι μόνο για τον τόπο αλλά για την ουσία αυτή εδώ τη συνεδρίαση. Ε, επίσης, θέλω να σας ευχαριστήσω ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, και κυρίως την εισηγήτρια την κυρία Στρίφερ αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως και την Λιθουανική Προεδρία για το επικοδομητικό έργο που διατέλεσαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων τριλόγου σχετικά με τον κανονισμό για τους Ευρωπαίους εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας. Αποτελεί μεγάλη τιμή για την ελληνική Προεδρία η ελληνική αυτή πρωτοβουλία του 2003 να ολοκληρώσει την νομοθετική της διαδικασία κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας. Στο πλαίσιο αυτό προσβλέπουμε σε θετική ψήφο από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι οι Ευρωπαίοι εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας πέραν του ότι αποτελούν καινοτομία σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η υποστηρικτική τους συνδρομή θα είναι καθοριστική σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παρόχου ανθρωπιστικής βοήθειας ανά την Ιφίλιο. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι η Ελληνική Προεδρία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να διοργανώσει η μερίδα σχετικά με την αξιολόγηση αναγκών, needs assessments, των φορέων αποστολή και υποδοχή εθελοντών ανθρωπικής βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό πρόκειται να γίνει τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο ε, του 2014. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Grazie Vice Ministro Gerentopoulos. Nel corso di questi sei mesi Ελπίζουμε του μήνε τη ελληνική Προεδρία ε, να έχουμε πραγματικά στενή συνεργασία. Α, Yes. Ε, ε, ε, εγώ ζητώ συγγνώμη. Επειδή τέθηκε και το θέμα της Συρίας, η συριακή ανθρωπιστική κρίση εντάσσεται στις άμεσες προτεραιότητες της ελληνική Προεδρίας, το είπαμε από την πρώτη στιγμή αυτό, δεδομένου ότι η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται. Εκεί πρόκειται για μια ανθρωπιστική κρίση η οποία έχει ξεπεράσει κάθε, κάθε φόβο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και τα κράτη-μέλη αποτελούν το μεγαλύτερο διεθνή δωρητή βοήθειας προς ανακούφιση των πληγένων από τη Συριακή κρίση. Η συνολική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιτροπή και κράτη-μέλη για ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά προγράμματα τόσο στη Συρία όσο και στις γειτονικές χώρες ξεπέρασε τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έως και το Δεκέμβριο του 2013. Την περασμένη εβδομάδα στη Διεθνή Διάσκεψη Δωρητών του Κουβέιτ 2, η Επίτροπος κ. Γεωργίευα ανακοίνωσε ότι από τον προπολογισμό της Επιτροπής 100 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 165 εκατομμύρια ε, δολάρια, εντός του 2014 ε, ε, πρόκειται να δοθούν και τα κράτη-μέλη ανακοίνωσαν ότι θα, θα, χορηγήσουν ανθρωπιστική και αναψυγιακή βοήθεια που ανέρχεται συνολικά σε 590 ε, εκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Τούτο σημαίνει ότι η χρηματοδότησή μας φτάνει πλέον τα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών από την αρχή της κρίσης. Ως Προεδρία του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στηρίξουμε στεναρά τη διεθνή πρωτοβουλία No Lost Generation που στοχεύει στην προστασία, την εκπαίδευση και την ψυχολογική στήριξη της Συριακής νεολαίας για να αποφύγουμε μελλοντικά ένα νέο ε, κύκλο βίας, μίσους και μεσηλοδοξίας σε μια περιοχή που έχει υποφέρει πάρα πολύ τις τελευταίες δεκαετίες. Εν ώψη δε της διάσκεψης Κουβέιτ 2 και στο πλαίσιο της ε, ομάδας εργασίας του Βουλίου Κοχάφα, η Ελληνική Προεδρία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γραμματεία του Συμβουλίου προετοίμασε κείμενο κοινών μηνυμάτων της Ένωσης το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση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 ε, χαρούμενοι για την δυνατότητα που έχουμε να συνεργαστούμε και προσβλέπουμε σε πολύ στενή συνεργασία ε, για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία για το εξάμεινο της Ελληνικής Προεδρίας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να είστε καλά.